Benvenuti a tutti. Καλώς ήρθατε όλοι. Καθίστε. Έχουμε δύο μέρες μπροστά μας, δύο μέρες ε, με πάρα πολλή δουλειά και θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη και εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Επίσης υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ τους διερμηνείς λέει ο πρόεδρος. Έγκριση των πρακτικών ε, των συνεδριάσεων της 22ης και 23ης Φεβρουαρίου. Άμα δεν έχουμε παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τότε θεωρείται εγκεκριμένη, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Η σημερινή συνεδρίαση έχει δορυφορική μετάδοση. Σας πληροφορώ επίσης ότι η συνεδρίαση αύριο το απόγευμα όταν ε, μαζί με τον George Lyon ε, θα παρουσιάσουμε τις σκέψεις ε, για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠΑ θα γίνει στην αίθουσα 2 του 2 και όχι σε αυτή την αίθουσα. Ξεκινάει λοιπόν η συνεδρίαση της Επιτροπής μας και θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης το νέο σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης μετά το 2013, νέα προσέγγιση και νέοι στόχοι. Κατόπιν ετήματος των συντονιστών, ανετέφει μία μελέτη για το θέμα ώστε να εμβαθυνθούν τα σχετικά με την ΚΑΠ μετά το 2013. ορίζω τον κύριο Ζων Κριστόφ Μπιγό, ο οποίος είναι συντονιστής και συντάκτης του, της μελέτης. Και ο κύριος Μπιγό θα μας κάνει μία παρουσίαση και μετά θα απαντήσει και στις ερωτήσεις μας. Χαιρετίζω και την εκπρόσωπο της Κομισιόν και δίνω το λόγο στον κύριο Μπιωγό για να μας παρουσιάσει την μελέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η, τη μελέτη που θα παρουσιάσω στα γαλλικά θα την δείτε σε διαφάνειες στα αγγλικά. Την μελέτη την έχουμε σε μία προσωρινή της έκδοση στο τραπέζι σας και σας παρακαλώ να μας ε, συγχωρέσετε. Πρόκειται για μία προσωρινή μελέτη με πολλά τυπογραφικά λάθη και προβλήματα συμβατότητας μεταξύ του κειμένου και του πίνακα. Θα έχετε την τελική έκδοση στην την επόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μία μελέτη που συνέταξαν οι οικονομολόγοι από 8 διαφορετικά κράτη και μας ζητήθηκε να γίνει ένας απολογισμός του συστήματος άμεσων πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ζητήθηκε επίσης να εξετάσουμε τις διάφορες ε, κριτικές ε, και μεταρρυθμίσεις που πρότειναν οι κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, τα κράτη-μέλη, αγροτικές οργανώσεις, δίνοντας και αριθμητικά στοιχεία για αυτές τις προτάσεις. Και μας ζητήθηκε επίσης να δούμε πώς θα λειτουργούσε η ενιαία ενίσχυση μετά το 2013. Στο, σε ένα πρώτο τμήμα της μελέτης θέλαμε να περιγράψουμε την τωρινή κατάσταση των άμεσων ενισχύσεων μετά από αυτόν τον απολογισμό που επιφέρει πολλές αλλαγές. Διευκρινίζω τι είναι το Single Payment Schemes SPS είναι η ενιαία ενίσχυση στα παλιά κράτη-μέλη και έχουμε το Single Era Payment Scheme στα νέα κράτη-μέλη. Χρησιμοποιώντας μικροοικονομικά και μακροοικονομικά στοιχεία, εξετάσαμε το πώς εφαρμόζεται το σύστημα στα διάφορα κράτη-μέλη για να απλουστεύσουμε εν ώψη του 2013 και μετά τις μεταρρυθμίσεις για τον απολογισμό. Είδαμε το πώς θα έχουμε τις ενιαίες ενισχύσεις, πώς διαμορφώνονται οι ενιαίες ενισχύσεις μετά από το 2013, εκτός από ορισμένες ζωοτροφές και το βαμβάκι. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια τεράστια ευελιξία για την κατανομή των πληρωμών, είτε το ιστορικό μοντέλο δηλαδή είτε άλλο, αλλά πώς αν πάρουμε το συγκεκριμένο κονδύλιο το δίνουμε σε άλλες πολιτικές. Ο διαχωρισμός δηλαδή μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ είναι ένας ε, τεχνητός διαχωρισμός και η γεωργική πολιτική υπόκειται αρκετά, σε μεγάλο βαθμό στην επικουρικότητα. Έχουμε το άρθρο 68 αλλά έχουμε ακόμη καμιά δεκαριά άρθρα που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν προπολογισμό από τον πρώτο πυλώνα αλλού. Όπως ας πούμε δράσεις για το περιβάλλον που εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα. Πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό και άμα δω την περίπτωση της Γαλλίας στα 5,6 δις ε, άμεσων ενισχύσεων αν η Γαλλία είχε χρησιμοποιήσει όλα τα συστήματα ευελιξίας θα είχε χρησιμοποιήσει 3,6 δις, πάνω δηλαδή από το μισό, όπως θα ήθελε. Αυτό είναι λοιπόν πολύ σημαντικό διότι δεν είναι σαφές το όριο μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληρωμών και θελήσαμε να δούμε συνολικά το σύστημα των ενιαίων ενισχύσεων στους διάφορους πυλώνες. Βλέπουμε ότι το, το γεωργικό εισόδημα εξαρτάται άμεσα από τις ενιαίες ενισχύσεις, ακόμη και σε, μία, μια μέτρια χρονιά όπως είναι το 2006 ή μια κακή χρονιά όπως το 2009. Με διακυμάνσεις ε, μεταξύ των κρατών μελών βλέπουμε η πληρωμή να μην είναι ένα τόσο σημαντικό ποσοστό στην αξία παραγωγής για την Ολλανδία ενώ είναι, είναι μεγάλο ποσοστό για την Φιλανδία και υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ γεωργών, παραγωγών και περιφερειών είτε πρόκειται για ενίσχυση ανεκτάριο ή αναεργαζόμενο. Μετά εξετάσαμε και τις διάφορες ε, κριτικές στο σύστημα άμεσων ενισχύσεων μετά από την μεταρρύθμιση του 2003 και μετά τον απολογισμό. Ορισμένες κριτικές μας φάνηκαν ε, άστοχες, αλλά άλλε ε, θεωρήσαμε ότι ήταν αρκετά σοβαρέ για να τις λάβουμε υπόψη μα όταν θα έχουμε ένα σύστημα άμεσων ενισχύσεων. Δηλαδή άνηση κατανομή αυτών των ενισχύσεων που σε ορισμένα κράτη-μέλη αντικατοπτρίζουν το, το παρόν και το παρελθόν. Έχουμε μετά ε, κατανομή ανάλογα με το ενεργητικό, δηλαδή πληρώνεται η γη, οπότε έχουμε διαφυγή εκτός γεωργικού τομέα και επίσης η cross compliance ε, που θα έπρεπε να, αφιερώνεται στο, να πηγαίνει στο περιβάλλον ε, δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά όλα αυτά τα στοιχεία στο μέλλον. Εξετάσαμε μετά τις προτάσεις που έγιναν και από βουλευτές για τη μεταρρύθμιση των άμεσων ενισχύσεων ή γενικότερα της ΚΑΠ μετά το 2013 και έχουμε πάνω από 40 προτάσεις πολύ λογικές που δημοσιεύθηκαν και που προβάλλονται από τα κράτη-μέλη, από γεωργικούς συνεταιρισμούς, από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή από think tanks. Μεταξύ αυτών των προτάσεων υπάρχουν πολλές διαφορές. Έχουμε προτάσεις για να καταργηθούν εντελώς οι ενισχύσεις της ΚΑΠ και άλλες προτάσεις να διατηρηθούν όπως έχουν ή να, να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα είναι αντισταθμιστικό λόγω των επιπλέον υποχρεώσεων που απαιτούνται από τους Ευρωπαίους γεωργούς λόγω του ανταγωνισμού ή λόγω των κοινωνικών διεκδικήσεων για την ευημερία των ζώων ή για τη χρήση ε, γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Μεταρρύθμιση λοιπόν του συστήματος σε ένα αντικυκλικό σύστημα ανάλογα με την κατάσταση των αγορών ή άλλες προτάσεις που αφορούν ε, στη χρήση του τωρινού προϋπολογισμού του πρώτου πυλώνα για να ε, δημιουργηθεί μία αμοιβή για τις υπηρεσίες που οι γεωργοί παρέχουν στην κοινωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι προτάσεις έρχονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις και έχουν εγκριθεί από άλλες οργανώσεις γεωκτημόνων, γεωργικών συνεταιρισμών ή κυβερνήσεων. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν συγκλήσεις στις τελευταίες προτάσεις που έγιναν Υπάρχουν όμως ε, μεγάλες διαφορές μεταξύ των ε, παρεμβαίνοντων είτε στον προπολογισμό μεταξύ κρατών μελών, στο επίπεδο των ενισχύσεων ή στο κατά πόσο θα πρέπει να συγχρηματοδοτούνται αυτές οι ενισχύσεις με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και εδώ υπάρχουν και μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των προτάσεων. Αυτές οι προτάσεις μας οδηγούν στο να διαπιστώνουμε ε, ορισμένες αρχές για να προτείνουμε ανατολισμό των ε, μελλοντικών καταβολών. Βέβαια, εμείς ε, θεωρήσαμε ότι εδώ ξεπερνιόνται τα όρια των αρμοδιοτήτων μας ως τεχνικών, δηλαδή να μπούμε εμείς στο πετσί των πολιτικών, πράγμα το οποίο δεν μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα. Και να προσανατολίσουμε τις ε, τωρινές καταβολές ε, προς ε, πολιτικές για το κοινό καλό, δηλαδή είτε τη δημόσια υγεία, είτε το περιβάλλον, είτε την ύπεθρο. Να μπορέσουμε δηλαδή να προστατεύσουμε το νερό, το περιβάλλοντα χώρο και ό,τι διαφυλάσσει το μέλλον της γεωργικής δραστηριότητας για το, το τωρινό σύστημα όπου έχουμε έναν πυλώνα χρηματοδοτούμενο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και έναν δεύτερο πυλώνα συγχρηματοδοτούμενο με τους εθνικούς προϋπολογισμούς οδηγεί σε μία αδιαφορία για την ε, χρηματοδότηση πολιτικών που αφορούν ε, τα κοινά αγαθά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι σε όλους τους πυλώνες θα πρέπει να υπάρχει μία συγχρηματοδότηση. Αυτό δημιουργεί θεσμικά προβλήματα σε επίπεδο προϋπολογισμού και ευρωπαϊκών αποφάσεων. Κοιτώντας τώρα τις επιπτώσεις ε, στα μικροοικονομικά στοιχεία και στο δίκτυο των λογιστικών πληροφοριών οι, τωρινές, οι τωρινοί κανόνες οδηγούν σε πολύ σοβαρές μεταφορές ε, μέσα στα κράτη-μέλη, ακόμη και αν κρατούσαμε σταθερούς τους δημοσιονομικούς φακέλους και πάντοτε με κριτήρια τα οποία δεν είναι πάντοτε αυτονόητα και χρειάζεται, απαιτείται μάλλον όλο ένα μεγαλύτερη επικουρικότητα για τον καθορισμό των κριτηρίων και την κατανομή των κονδυλίων αλλά με κοινού κανόνες ούτως ώστε να αποφύγουμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τις μεταρρυθμίσεις ε, του συστήματος άμεσων ενισχύσεων προτείναμε, αλλά ξεφεύγοντας πάντοτε από το πεδίο της τεχνικής ε, πραγματο στα πλαίσια του κονσόρσιουμ όπου συμμετείχαν 15 οικονομολόγοι από διαφορετικές χώρες και που διαφωνούσαν σημαντικά ως προς το βαθμό ε, συγχρηματοδότησης ε, ή δημοσίων επενδύσεων κλπ. Φαντάζομαι βέβαια ότι οι διαφωνίες που είχαμε εμείς ε, στο δικό μας κονσόρσιουμ θα είναι μπορούν να θεωρηθούν ε, μηδενικέ ε, εν ώψη των διαφωνιών που θα υπάρχουν σε πολιτικό επίπεδο. Θεωρήθηκε ότι άμεσες ενισχύσεις, η ενιαία η μοναδική μάλλον η ενιαία πληρωμή δεν θα πρέπει να καταργηθεί, θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδος και άμα κάτι τέτοιο συμβεί θα πρέπει να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και μακρύ αλλά και σαφέστατο ούτως ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να το καταλαβαίνουν και οι παραγωγοί χρειάζονται και μία συνάφεια και άμα πάρουμε το παράδειγμα των νέων κρατών μελών όπου έχουμε τις πληρωμές πάντα σε μεταβατική περίοδο και για δύο κράτη-μέλη θα αυξάνονται μέχρι το 2016 φαίνεται σαφώς ότι το να αυξήσουμε αυτές τις ενισχύσεις για να τις κόψουμε μετά μαχαίρι δεν έχει νόημα. Χρειάζεται όμως ένας επαναπροσανατολισμός του τωρινού συστήματος για χρηματοδότηση δημοσίων αγαθών που σήμερα δεν πληρώνονται από την αγορά, από την αγορά. τοπίο, ε, βιοπικιλότητα, περιβάλλον, ύπεθρος. Πρέπει λοιπόν εμείς ε, να, οδηγεί, προχωρήσουμε το σύστημα πρικοδοτώντας με κονδύλια για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τους στόχους και αν δεν υποστηριχ... υποστηρίζεται Συγγνώμη, αν δεν ακολουθείτε με αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, τότε οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να μειωθούν. Τώρα, για τον δεύτερο πυλώνα υπάρχει ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, Σίγουρα δεν θα πρέπει να συγχωνευτεί, αλλά ορισμένα ε, σχήματα τύπου ενίσχυση μειονεκτικών περιφερειών θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν μέσα σε μια γενικότερη βεντάλια περιφερειακών πληρωμών ή σε ένα ποσοστό ενισχύσεων ανεκτάριων στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα. Να υπάρξει δηλαδή μια ομαδοποίηση ορισμένων καταβολών που έχουμε στους δύο πυλώνες. Λοιπόν, θέλουμε να προχωρήσουμε προς ένα σύστημα πιο ομοιογενές με λιγότερες ανισότητες μεταξύ περιφερειών και γεωργών και οι προσωμιώσεις που κάναμε είναι πραγματικά ε, συγκλονιστικές. Βλέπουμε εμείς μέσα από αυτές τις προσωμιώσεις ότι δεν τίνουμε πράντα προς την αρχική μας κατεύθυνση. Όταν πληρώνουμε εμείς ανά εργαζόμενο μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερα στρεβλωμένα αποτελέσματα αντίθετα από ό,τι φανταζόμασταν. Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε μεταφορές από ζώνες εντατικής ε, κτηνοτροφίας ε, μπορούμε να, μπορεί να έχουμε μεταφορά προς ε, ε, αμπελουργία ψηλής ποιότητας. Αν αποφασίσουμε νέους κανόνες λοιπόν πληρωμής θα πρέπει να έχουμε κανόνες ακριβέστατους για να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι οποίες δεν είναι καθόλου μα καθόλου αυτονόητες. Επίσης ε, μια μεγάλη επικουρικότητα ούτως ώστε να αποφευχθούν όλα αυτά τα στρεβλά φαινόμενα γιατί τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες είναι οι πιο αρμόδιοι να ξέρουν ποια είναι η αποτελεσματικότητα των πληρωμών. Τώρα πολλές κοινωνικές ομάδες, π.χ. οι συνεταιρισμοί και ορισμένα κράτη-μέλη μας ζήτησαν να έχουμε μια ε, προσαρμογή στον τιμάριθμο αυτών των ενισχύσεων ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις γεωργικές τιμές. Εμείς θεωρήσαμε όμως ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε στρεβλώσεις και μπορώ να απαντήσω σε αυτό στις ερωτήσεις. Μία δεύτερη συνιστόσα, πέρα από την εισοδηματική ενίσχυση, δηλαδή την ενίσχυση των δημοσίων αγαθών, θέλει να αποφύγει, να αποφύγει τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα που έχουμε στον δεύτερο πυλώνα, ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο στοιχίζει ακριβά από διοικητικής πλευράς. Προξενεί και δυσκολίε στην εφαρμογή σε ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν μεγάλο πληθυσμό μικρών γεωργών, μικρών εκμεταλλεύσεων δηλαδή και προσπαθούμε στηριζόμενοι και στις εργασίες που ήδη έχουν υλοποιηθεί ως προς το τα δημόσια αγαθά να προτείνουμε κάποιες ε, ιδέες για στήριξη, για αποζημίωση για την παροχή δημοσίων αγαθών σε ε, καταρχάς καταποκοπήν σύστημα, κάπως περιφερειοποιημένο, αλλά και στη συνέχεια πιο στοχευμένο, αντίστοιχο με αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ως προς τα μέτρα τα αγροπεριβαλλοντικά. Agri-Environmental Schemes. Και έτσι αφήνουμε αρκετά ευρύ περιθώριο και για την επικουρικότητα και στο θέμα αυτό για τα κράτη-μέλη. πρωταρχικές συνέπειες. Καταρχάς έχουμε μια πιο ομοιογενή κατανομή των ενισχύσεων όσο διατηρείται η ενίσχυση στο εισόδημα τουλάχιστον, διότι εδώ πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ε, και να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό μας επιτρέπει η κατάσταση της αγοράς με ποια ταχύτητα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο σύστημα δημοσίων ενισχύσεων, οι προλογισμοί πάνω απ' όλα τι επιτρέπουν, σε ένα σύστημα λοιπόν στο δυνατόν πιο ομοιόμορφο με μία ενίσχυση ενιαία κατά, κατά πάσα πιθανότητα αναεκτάριο και με ένα ταμείο για το εργατικό δυναμικό. Αυτό θα είναι το λιγότερο κακό μέτρο από την άμεση δηλαδή ενίσχυση για το εργατικό δυναμικό ανεργαζόμενο, ένα σύστημα το οποίο με τις προσωμιώσεις μας φάνηκε να προξενεί δυσκολίες. Ένα άλλο ε, δεδομένο, μια άλλη συνέπεια θα ήταν οι μεταφορές, η πιθανότητα μεταφορών, η μετακίνησης από, ε, μεταξύ κρατών μελών με μια ενιαία δηλαδή πληρωμή ένα εκτάριο, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι θα μπορούσαν οι ενισχύσεις να ε, λάβουν υπόψη την αγοραστική δύναμη σε ευρώ μέσα στο κάθε κράτο μέλο, τι διαφορέ δηλαδή σε αγοραστική δύναμη, αλλά και πάλι αυτές τις δημοσιονομικέ ε, μεταφορέ θα πρέπει να τι εξετάσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μαζί με τα διαφορετικά ταμεία, μαζί με τι εκπτώσεις κτλ. Και ενδεχομένω, θα ήταν και χρήσιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο να προσδιοριστεί ένα πακέτο εθνικό με βάση σχετικά αντικειμενικά κριτήρια, ανακράτο δηλαδή. Ε, ε επιφάνεια γεωργικών ε, γεών, εργατικό δυναμικό, ε, εκτάσει υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και ούτω καθεξή με τέτοια κριτήρια. Και μέσα σε αυτό το πακέτο, το, το εθνικό, να αφήνουμε μεγαλύτερο περιθώριο για την επικουρικότητα. Για τη συγχρηματοδότηση. Χρήσιμο μας φαίνεται να προχωρήσουμε προς μια συγχρηματοδότηση ανάλογη λίγο πολύ με, αυτό, με αυτή την οποία να εξασφαλίσουμε τους δύο πυλώνες αυτή τη στιγμή, έστω και αν μπορεί η περίμετρος αυτών των δύο πυλώνων να τροποποιηθεί. Το πρόβλημα βεβαίως θα είναι η μετάβαση. Και το πώς θα διαχειριστούμε δηλαδή τη μετάβαση. Και επίση, αν υπάρχει και εθνική συγχρηματοδότηση, πράγμα το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα και εθελοντική ε, χρηματοδότηση κονδύλια επιπλέον, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε σημαντικέ ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να σταθμίσουμε λαμβάνοντα υπόψη ή ε, εισάγοντα κάποια ε, διαφορετικά ποσοστά χρηματοδότηση, πάλι στηριζόμενα αντικειμενικά κατά το δυνατόν κριτήρια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η εισαγωγή πολιτικών με εθνικό χαρακτήρα. Βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε και να διατηρηθεί ένα κοινό πλαίσιο. Ένα πραγματικά ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κοινή πολιτική που θα έχει την πτυχή του δημόσιου αγαθού ε, έτσι ώστε να αποφεύγονται ειδικά στον τομέα αυτών οι στρεβλώσει του ανταγωνισμού και όπου θα υπάρχει και ένα σαφέστατο ορισμό, ενιαίο ορισμό ω προ το σημείο αναφορά. Δηλαδή, τι θα ζητούμε από το γεωργό ποια κριτήρια θα του απαιτούμε να τηρεί. Περιβαλλοντικά, ε, κτηνοτροφικά, προστασία του τοπίου και χάρη στα οποία θα μπορεί να διεκδικεί επιπλέον πληρωμές υπό την έννοια του δημοσίου αγαθού. Αφού ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπονται κάποια ελάχιστα κριτήρια, αρκετά διαφορετικά μεταξύ των κρατών μελών, για να δώσω ένα παράδειγμα την ε, ε, ευημερία των ζώων, στις, στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία, οι προδιαγραφές σχετικές με την προστασία των ζώων και την ευημερία τους είναι υψηλότερες. Άρα εκεί μπορεί ένας γεωργός, ένας κτηνοτρόφο καλύτερα, να έχει τη σχετική ενίσχυση προκειμένου να εξασφαλίσει επίπεδα προστασίας τα οποία για τα άλλα κρατημέλη δεν του προσφέρουν τέτοια οικονομική ενίσχυση και έτσι θα έχουμε στο τέλος ε, στρεβλώσεις μη επιθυμητές φυσικά. Τώρα, ε, η συμβατότητα των διατάξεων αυτών περί των ε, κρατικών ενισχύσεων, των δημόσιων ενισχύσεων, σε σχέση με του διεθνεί κανόνε, την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου ιδιαίτερω, δεν βλέπουμε ιδιαίτερο πρόβλημα ε, και μάλιστα εάν αποφασιστεί η εισαγωγή ενό αντικυκλικού αντικυκλικής συνιστώση, πράγμα το οποίο δεν θα προτιμούσαμε εμεί, δεν θα συνιστούσαμε εμεί, ίσω χρειαστεί να λειτουργήσει το κριτήριο του ε, το συνολικό λεγόμενο κριτήριο στρέβλωσης του ανταγωνισμού της Δόχα ε, overall distortion ε, system και εκεί θα χρειαστεί περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εισαχθεί αυτό το κυκλικό σύστημα. Για δε τις σχέσεις με τις αγορές. Ένα σύστημα άμεσων ενισχύσεων, έστω και αναθεωρημένο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη ρύθμισης των αγορών. Η ρύθμιση η οποία θα έχει σαν στόχο και να αντιμετωπίσει την μεγάλη πτυτικότητα των εσόδων και των αμοιβών στον τομέα αυτών που είναι απαραίτητη. Ασφαλώς μπορούν να διαδραματίσουν οι ε, καταβολές ε, δημόσιου χρήματος σταθεροποιητικό ρόλο, το έχουμε ήδη δει αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να έχει κανεί ταμπού, οι, πληρω... οι καταβολές δηλαδή αυτών των ενισχύσεων μπορούν να συνδυαστούν, να συνδεθούν δηλαδή με την παραγωγή εφόσον αυτή ε, εξεταστεί υπό το πρίσμα του δημόσιου αγαθού, φερρυπίν, κτηνοτροφία σε απομακρυσμένες περιοχές, περιφερειακέ περιοχέ, και άρα μπορούμε να δούμε εκεί πέρα την ενεργοποίηση του άρθρου 68. Πλην όμω το σύστημα των άμεσων πληρωμών δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πιο παραδοσιακή κοινή γεωργική πολιτική, δηλαδή τη ρύθμιση των αγορών. Για τα τελικά συμπεράσματα. Υπάρχουν ασφαλώς θεσμικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν από την επιβολή ενός νέου συστήματος στο μέλλον Συστήματο πληρωμών, δηλαδή κυρίως ε, με βάση τα όσα προτείνουμε εμεί δηλαδή ενίσχυση τη συγχρηματοδότησης, διεύρυνση της συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των διακρίσεων ε, εν ώψη του δεύτερου πυλώνα με το τωρινό σύστημα, επιπλέον προστασία, ενίσχυση προστασία των δημοσίων αγαθών και δεδομένου ότι ε, αυτό που προτείνουμε εμεί είναι τα κράτη-μέλη που τώρα έχουν μεγάλη ετερογένεια προ τι δομέ του να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν κατά το δοκούν και κατά τι ε, τοπικέ του ανάγκε το σύστημα, ε, αλλά παράλληλα πρέπει να τηρούνται και κάποιοι κοινοί κανόνε σε κοινοτικό επίπεδο και για την στήριξη του εισοδήματο, αλλά και στην λεγόμενη συνιστόσα των δημοσίων αγαθών. Θα πρέπει εδώ να δούμε ένα σύστημα αρκετά πιο περίπλοκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Ζαν Κριστόφ Μπυρό. Μας δώσετε μερικά πολύ σημαντικά στοιχεία. Οι συναδελφοί ήδη έχουν ζητήσει το λόγο. Αρχίζουμε με τον κύριο Παπαστάμκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μπυρό και στο πρόσωπό του τους ε, συντάκτες ε, αυτής της μελέτης, η οποία πράγματι είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το έργο το οποίο επιτελούμε. Ε, βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, ε, θα ήθελα να δω σε κάθε σενάριο εναλλακτικό πρέπει να δούμε και την δημοσιονομική αναφορά. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αυτό, ούτως ώστε να έχουμε και ένα επιστικό επιχείρημα και απέναντι στους αγρότες των χωρών μελών τους οποίους εκπροσωπούμε, αλλά και σε όσους προβάλλουν ενστάσεις για το ύψος του προϋπολογισμού που κατευθύνεται στη Γεωργία. Ε, νομίζω ότι τότε μια μελέτη θα διεκδικούσε πραγματική πληρότητα. Κατά την προσωπική μου γνώμη, οι άμεσε ενισχύσει πρέπει να σταθούν πάρα πολύ σοβαρά στο θέμα των αμέσων ενισχύσεων, γιατί είναι, αυτές, είναι αυτό το εργαλείο που συγκρατεί τον πληθυσμό στην ε, ευρωπαϊκή ύπεθρο ε, και κακά τα ψέματα αποτελεί και κίνητρο για τη συνέχιση της γεωργικής παραγωγής. Βεβαίως το, ερώτημα της ε, δίκαιης κατανομής των ενισχύσεων, σε ποιους θα κατευθύνονται οι ενισχύσεις και με ποια κριτήρια θα κατανέμονται, παραμένει κρίσιμο κατά τη γνώμη μου. Ε, ένα ερώτημα που θα ήθελα να θέσω στον κύριο Μπυρό, το, το υπενήχθηκε, αλλά αν μπορούσε να μας φωτίσει λίγο περισσότερο, εάν το θέμα της συγχρηματοδότησης του πρώτου πυλώνα είναι συμβατό με την ε, κοινοτική νομοθεσία, με το το νομικό instrumentarium της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής όπως ισχύει και επίσης θα ήθελα να δω την έκθεση να συμπληρώνεται με τις επιπτώσεις όλης της συζήτηση για την μετά το 2013 κοινή αγροτική πολιτική στις, στη γεωργία μικρής κλίμακας. Αν η γεωργία μικρής κλίμακας, η οποία συνδέεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ήπεθρο, εάν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ερευνητικό σημείο αναζήτησης και επεξεργασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Παπαστάμκο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. James Nicholson. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση υποθέτω σε κάθε χώρα μέλος η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο καθένας γνωρίζει καλύτερα την κατάσταση στη χώρα του. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται σε όλες τις 27 άλλες χώρες. Η έκθεση του κ. Λάιονς πολύ σωστά επεσήμανε ότι υπάρχει τεράστια ανισότητα στην ε, κατανομή πόρων μεταξύ κρατών μελών. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Το σύστημα αυτό των ενιαίων πληρωμών σε... είναι σημαντικό προκειμένου να συνεχίσουν να επιζούν μικρές οικογενειακές γεωργικές μονάδες και στο μέλλον. Ίσως κάτι δεν κατάλαβα καλά, ίσως είπατε και δεν το κατάλαβα καλά. Όταν ε, συνδέσαμε με το check-up, το, την ενιαία πληρωμή, είχαμε στοιχεία σχετικά με το τι ζωικό κεφάλαιο Φερρυπίν ε, στην παραγωγή ε, προβάτων, προβατίνες κλπ. Κι αν υπήρξε μείωση σε περιοχές ευαίσθητες όσον αφορά, όσον αφορά το περιβάλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρειαζόμαστε απάντηση πριν δούμε πώς θα γίνει η διανομή των κονδυλίων. Γιατί οι περισσότεροι γεωργοί, μερικοί αποσυνδέουν περισσότεροι από άλλους, αλλά μερικά συστήματα στηρίζονται στο τύχη στο αγρόκτημα του 2000-2001 και μετά το 2013 φυσικά αυτό δεν θα είναι αποδεκτό. Άρα οι αλλαγές που θα γίνουν θα πρέπει να είναι ελεγχόμενες. Συγχρηματοδότηση. Αν, δεν, αν πάψει να είναι υποχρεωτικός ο κανόνας αυτός και γίνει προαιρετικός τότε από την κοινή γεωργική πολιτική μήπως θα φύγει το κοινό ή θα έπρεπε να φύγει το κοινό, δεν θα έχουμε πια κοινή πολιτική γιατί κάθε χώρα ανάλογα με, το, με τον τρόπο της θα το αλλάζει το σύστημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε Τζέιμς. Ε, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Άλμπερτ Τες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον συντάξη της εκθεσής. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τόσο μας είπε. Αν και θεωρώ ότι χρειάζονται και κάποιες ε, προσθήκες. Ο πρώτος πυλώνας πιστεύω θα πρέπει και στο μέλλον να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς συγχρηματοδότηση. Τον χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την ε, σύντηση, τη διατροφή δηλαδή 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης. Ο πρώτος λοιπόν πυλώνας θα πρέπει και μετά το 2013 να συνεχίσω, όχι όμως με την, ε, με την ίδια, ε, στο ίδιο μέγεθος. Έτσι λοιπόν, όταν ε, απαιτεί η Διεθνής Οργάνωση Εμπορίου οι πολύ ψηλές προδιαγραφές από την Ευρώπη, θα είμαστε σε θέση να ε, στηρίξουμε τους αγρότες μας ε, στις περιοχές οι οποίες έχουν περισσότερες δυσκολίες και να αιτιολογήσουμε τη στήριξη αυτή με σοσιαλιστικές πληρωμές από τον πρώτο πυλώνα. Για δε το δεύτερο πυλώνα που λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει σε ένα κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότηση, αυτό θα μπορούσαμε και να το συζητήσουμε. Αγαπητέ κύριε Παπαστάμκο, ε, θα μπορούσα να διαπιστώσω μια κάποια διαφοροποίηση ως προς τις δικές μου θέσεις, διότι στο δεύτερο πυλώνα ε, λέτε θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 25% ε, συγχρηματοδότηση και θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και το 50% της συγχρηματοδότησης. Αυτό θα μπορούσαμε να το δεχθούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα ιδιαίτερη στρέβλωση ανταγωνισμού. Αλλά το δεύτερο πυλώνα πάνω απ' όλα τον χρειαζόμαστε για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, ε, γεωργική αναμετατροπή για την υποστήριξη των ε, πιο δύσκολων περιοχών, των ορεινών περιοχών με τις ισοσκελιστικές εξωτικές δηλαδή πληρωμές. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μόλις ξεκινάει. Τον επόμενο μήνα θα έχουμε την ευκαιρία πολύ πιο διεξοδικά να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι πάντως μια καλή βάση για συζήτηση αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση σχετικά με τα δημόσια αγαθά, διότι η έννοια δημόσιο αγαθό δεν έχει οριστεί. Έπειτα βλέπω ότι συχνά Ο όρος δημόσιο ή δημόσιο αγαθό χρησιμοποιείται κατά κάποιο τρόπο σε αντίθεση με τα γεωργικά προϊόντα, που είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Με βάση τις προβλέψεις των ΗΕ προβλέπεται αύξηση περίπου, θα πρέπει να έχουμε αύξηση 70% των, της γεωργικής παραγωγής, γιατί ο αριθμός των λιμοκτονούν ατόμων όλο και αυξάνεται. Το τρόφιμο λοιπόν θα πρέπει να θεωρείται ως ε, δημόσιο αγαθό παρκόμενο από τη Γεωργία. Ανιώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εφτά μικρά σχόλια. Ο μιλητής είπε να μείνουν μερικά ε, πληρωμές για τα μυρικαστικά ή τα χορτοφάγα Αυτό δεν το έχουμε στην Αγγλία. Υποθέτω υπάρχουν γεωργοί 50% του παλιού συντελεστή και την ε, κατά αποκοπή πληρωμή. Νομίζω αυτό το, αυτή η στρεβλή υποστήριξη δεν πρέπει να εξακολουθήσει. Επαναπατρισμό, μερικός επαναπατρισμός της ΚΑΠ. Επικίνδυνος. Πολλές κυβερνήσεις και οι δικοί μας το βλέπω σε έναν τρόπο να πάψουν να δίνουν χρήματα στους γεωργούς και να βρουν άλλους τρόπους και χρήση. Συμφωνώ ότι η χρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα είναι αγκαία. Ελπίζω αν και αναφέρθηκε στην έκθεση, πάντως στην, ε, στην οθόνη δεν το είδαμε, δηλαδή να ζητήσουμε από τους γεωργούς να πάρουν μέρος σε κάτι που δεν έχει αποδειχθεί αλλαγή για το κλίμα. Ελπίζω να μην ήταν στην παρουσίαση και να μην συνεχίσουμε να συζητάμε γι' αυτό. Τέσσερα. Είμαι κατά του πυλώνα 2, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα στην εκμετάλλευση, εκτός αν έχουμε πολύπλοκες μεθόδους και έχω κάνει ένα υπολογισμό κόστος στο παρελθόν. Υπάρχει μια εξαίρεση όμως, χρήματα του δεύτερου πυλώνα για να συμμορφώνονται οι γεωργοί με την κοινωτική νομοθεσία. Η γαλακτοπαραγωγή, η Φερρυπίν ή ακόμα και αυτοί που παράγουν πουλερικά και αυτοί το ίδιο πρόβλημα έχουν κατά κάποιο τρόπο. Σχόλιο 6. Δεν θέλω να μπει κανένα στοιχείο εργατικών στο θέμα αυτό. Φαντίστε, μια, ένα, μια εκμετάλλευση η οποία έχει γουρούνια, πουλερικά και θα υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν εκεί. Ο Γιώργο αυτό θα πάρει περισσότερα χρήματα, αλλά οι συνάδελφοί του, οι ανταγωνιστέ του, που δεν έχουν γη αρρώσιμη, όπω έχει αυτό στο παράδειγμα, θα πρέπει να τον ανταγωνιστούν με άλλου όρου. Και επιπλέον, όταν θα αρχίσουν τα σούπερ μάρκετ να βλέπουν ότι επιδοτούνται οι παραγωγοί πουλερικών, θα ρίξουν την τιμή που δίνουν. Τέλος δεν ακούσαμε τίποτα για το cross compliance η γενική φιλοσοφία τι είναι, ότι θα δυσκολέψουν τα πράγματα ή ότι θα διευκολυνθούν όσο προχωράμε στο μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Ανιώ, Μισελ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ το συντάκτη της εκθέσεως. Σημειώνω ότι στην αρχή της ομιλίας του υπογράμμισε ότι θα μπορέσουν στην προσεχή περίοδο οι γεωργοί της Ευρώπης παρόσα ορισμένοι προσπαθούν να υπονοήσουν να επιβιώσουν χωρίς τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων δηλαδή. Αναφερθήκατε σε διάφορες, σε διαφορετικές υποθέσεις δηλαδή, μιλήσατε για το εργατικό δυναμικό. Ε, με τις προσωμιώσεις λοιπόν ερωτώ εάν δοκιμάσατε το, ε, την προβολή της εισαγωγής της ενίας πληρωμής μέσα στην ενία μάλλον πληρωμή τις διάφορες επιβαρύνσεις που ισχύουν ανακράτος μέλος. Ο κύριος Καπούλα Muito obrigado. Eu quero agradecer este estudo, que é um excelente contributo para nós, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ το Στάκτη για την έκθεση αυτή. Είναι, πιστεύω, ξέρετε, συμβολή στις εργασίες μας συχνά ε, αναμειγνύεται η τεχνικού χαρακτήρα συζήτηση με την πολιτική. Βεβαίως κάθε πολιτική συζήτηση και απόφαση θα πρέπει να στηρίζεται σε, στα τεχνικά στοιχεία, στις τεχνικές γνώσεις. Αλλά το δεν θα πρέπει και να αντιστρέφουμε την κατάσταση. Αυτό λοιπόν το οποίο θα τώρα να πράξουμε είναι να συζητήσουμε ένα πρότυπο, μια, ένα σύστημα, ένα αρχιτεκτόνημα αν θέλετε για την γεωργία της Ευρώπης. Και άπαξ και προσδορίσουμε τη δομή αυτή που θέλουμε, θα βρούμε και την τεχνική στήριξη. Το πλεονέκτημα που μας προσφέρει αυτή η έκθεση είναι ότι μας δίνει κάποιες τεχνικές λύσεις εφαρμόσιμες και γι' αυτό την κρίνω θετικά την έκθεση. Είναι πολύ θετικό το να δούμε παραδείγμα ότι, ότι ε, η γραμμή αυτή Τη στις εκθέσεις συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με τις θέσεις της σοσιαλιστική ομάδας. Της ομάδας έχουμε υποστήριξη για τους ε, γεωργούς ανά εκτάριο μια ενίσχυση η οποία μπορεί να ε, αιτιολογηθεί και με τους όρους της διατήρησης θέσεων εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εκεί που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι στο να αντιληφθούμε πώς θα συνδέσουμε μεταξύ τους αυτές τις λύσεις. Έγινε λόγος για πρώτο πυλώνα, για δεύτερο πυλώνα, κάποιοι ήταν τελείω κατά του δεύτερου πυλώνα. Ο καλύτερος τρόπος να επιλύσουμε το πρόβλημα πιστεύω είναι να ξεφύγουμε από την λογική των δύο πυλώνων και να βρούμε ένα ενιαίο σύστημα πληρωμών, ένα σύστημα ενιαία πληρωμή, μάλλον, με βάση μια κοινή λογική, μια απλή λογική και όχι τα κριτήρια που είχαμε στο παρελθόν, γιατί από το 2003 και μετά έχουμε προχωρήσει από τα παλαιά παραδοσιακά κριτήρια. Ε, έτσι λοιπόν βλέπω να συζητείται το ζήτημα της συγχρηματοδότησης ως τεχνικό, ενώ είναι στην πραγματικότητα πολιτικό ζήτημα. Διότι άπαξ και αποφασίσουμε για το πρότυπο που θέλουμε, για το σύστημα που θέλουμε, και μόνο άπαξ το και το αποφασίσουμε αυτό θα μπορέσουμε να δούμε εάν επιθυμούμε τη συγχρηματοδότηση ο σύστημα ή όχι. Αυτή τη στιγμή που έχουν μεγάλα ε, ελλείμματα τα κράτη-μέλη και όπου η προτεραιότητά τους δεν εντοπίζεται στη γεωργία, η συγχρηματοδότηση θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ε, στρεβλώσεις της αγοράς και να αποβεί εις βάρος τελικά του κόσμου της γεωργίας στην Ευρώπη συνολικά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να κρίνουμε αργότερα δηλαδή. Αλλά πάντως η έκθεση είναι πολύ χρήσιμη και θα είναι πολύ χρήσιμη την ώρα που θα κληθούμε να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Ο κύριος Λάιν έχει το λόγο. George Λάιν. Θα ήθελα και εγώ πρόεδρε να πω δύο λόγια. Με κάλυψαν αρκετοί από τους προλαλήσαντες για την πρώτη μου παρατήρηση οι προτάσεις σας για τη συγχρηματοδότηση φαίνεται να ισοδυναμούν με την επανεθνικοποίηση τη κοινή γεωργική πολιτική. Πώ μπορεί να υπάρξει κοινή γεωργική πολιτική μετά από το τέλο αυτή τη διαδικασία, εάν ακολουθήσουμε τα όσα μα λέτε, ή στο μεγαλύτερο του βαθμό, εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, παρακαλώ, τι θα μείνει τελικά το κοινό σε αυτή την κοινή γεωργική πολιτική, εάν δεχθούμε τι δικέ σα προτάσει. Και δεύτερον, η συζήτηση σχετικά με το εργατικό δυναμικό και την υποστήριξή του και τα κριτήρια για την υποστήριξη αυτή. Και πάλι μιλούμε για σημαντική επανακατανομή της στήριξης των ενισχύσεων. Έτσι λοιπόν μπορεί και να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση ορισμένες, ορισμένα είδη παραγωγής, δηλαδή να στρεβλωθεί και πάλι ο ανταγωνισμό και δι τη ε, Ευρώπη συνολικά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορείτε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ, Μάρτιν Όσλινγκ. Για τη συγχρηματοδότηση, αυτό που θα πω εγώ μόνο είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος με τη συγχρηματοδότηση να βάλουμε και τα φόπλακα της γεωργικής πολιτικής, της κοινής γεωργικής πολιτικής, γιατί όπως τα ορισμένα κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτήσουν. Και γι' αυτό θα πρέπει πολλά από τα μέτρα του πρώτου πυλώνα να χαρακτηριστούν και να παραμείνουν ως ευρωπαϊκά μέτρα. Η έννοια των δημοσίων αγαθών βεβαίως θέλει πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό και περιγραφή. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής πρέπει επίσης να το λάβουμε υπόψη. Στον πρώτο πυλώνα όμως όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν και να τύχουν προστασίας. Το εργατικό δυναμικό. Μέχρι τώρα ε, βλέπω να αντιμετωπίζεται κάτι το αρνητικό. Δεν βλέπω δηλαδή που ε, επισημαίνετε εσείς τη δυνατότητα για βελτίωση των συνθήκων για το εργατικό δυναμικό. Η εντατικοποίηση είναι εκείνη η οποία έχει οδηγήσει στην ε, συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού και όχι η εκτακτικοποίηση. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να δώσουμε λίγο βάρος. Και επίσης θα πρέπει να διερωτηθούμε τι γίνεται σε σχέση με τους κανόνες των αγορών. Δεχόμαστε η γεωργία να λαμβάνει το 50% των, ε, του, του κοινοτικού προϋπολογισμού ακόμη και στο μέλλον. Είναι δυνατόν να διατηρήσουμε αυτή την ενίσχυση των εισοδημάτων και δεν θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σε ε, συνδυασμό όχι μόνο με τους κανόνες της πολιτικούς, πολιτικής αλλά και τις λειτουργίες των αγορών. Η κυρία Γκαρσία. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, παρουσίασή του, αλλά ανησυχώ για δύο πράγματα. Όταν ιδρύθηκε η ΚΑΠ στη συνθήκη της ε, Ρώμης, είχε ως στόχο την παραγωγή της τροφίμων σε... που εξασφαλίζει την αυτάρκεια στην Ευρώπη σε λογικές τιμές. Αν σταθούμε σε αυτήν, την αρχή τότε μπορούμε κάλλιστα να την καταργήσουμε. Αλλά σήμερα αν χρειάζεται μια κοινή πολιτική είναι αυτή η πολιτική η οποία έχει τεράστια προβλήματα σήμερα και λόγω της πολυεθνικότητας και ποικιλότητα του πληθυσμού στην Ευρώπη αλλά και της έλλειψης θέσεων απασχόλησης και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην πολιτική του 2013. Επίσης θα πρέπει να σταθούμε και σε άλλα στοιχεία όπως είναι προστασία ε, ε, του περιβάλλοντος όπως προστασία των εργασιακών κανόνων της ΔΟΕ. Και θα έπρεπε αυτό να το δούμε και στο γύρο της ΔΟΑ. Αν υπάρχει ένας κίνδυνος σήμερα για την ΚΑΠΕ είναι το εξωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που απογυμνώνει την ΚΑΠΕ σε πολλές ευκαιρίες θα ήθελα η μελέτη να δει και το θέμα του διεθνούς εμπορίου και το πώς επηρεάζει το διεθνές εμπόριο τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα. Επίσης, η παραγωγή είναι δύο τύπων. Είναι αφενός η γεωργή και η κτηνοτρόφη. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Ούτε οι εκμεταλλεύσεις τους, ούτε η δουλειά τους. Και θα έπρεπε να μην αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο ως προς τις ενισχύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να είστε πιο συγκεκριμένος αυτά. Ναι, δεν είχα καταλάβει Ευχαριστώ πολύ για τι ε, παρατηρήσει, για την επιστημονική μελέτη. Θα ήθελα να πόσο κάποιε σύντομε ερωτήσει, παύλα παρατηρήσει. Καταρχά, κάτι που δεν κατάλαβα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αφενός μεν το ζήτημα της ε, ε, αντιμετώπιση των διαφορών, αφετέρου δε την προσπάθεια να διατηρήσει μια κοινή πολιτική. Μια ενότητα δηλαδή. Αυτό το εξασφαλίζει ο πρώτος πυλώνας. Ενώ ο δεύτερος στόχο έχει να ε, εξασφαλίσει και να προσθέσει ενδεχομένω και τις ιδιαιτερότητες τις τοπικές. Θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να παραμείνουν οι δύο πυλώνες και για το μέλλον. Δεύτερο ερώτημα. Συγχρηματοδότηση. Αν σας κατάλαβα καλά, υποστηρίζετε ρητά την συγχρηματοδότηση, δηλαδή την κρίνετε θετικά. Έχετε κάποιες προτάσεις συγκεκριμένες για τα ποσοστά ε, στα οποία θα κρίνατε αποδεκτή τη συγχρηματοδότηση. 20, 25, 50, πόσο της εκατό. Τρίτο ερώτημα. Αντικίνητρα, λάθος κίνητρα. έχουμε ένα στόχο, επί παραδείγματι, να αντιμετωπίσουμε την έξοδο από το χώρο της υπαίθρου, την διαφυγή από την υπαίθρο του εργατικού δυναμικού. Τα προβλήματα αυτά που έχουμε σε σχέση με τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν οι πολιτικές οι οποίες έχουν, από ό,τι έχουμε ήδη διαπιστώσει, ε, προτείνει αντικίνητρα ουσιαστικά, δηλαδή αντιπαραγωγικά κίνητρα και αυτό το λέω εγώ γιατί από την πρώην λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας ε, είδα ενώ δεν υπάρχουν στην κοινοτροφία πολύ μεγάλε διαφορέ στι αμοιβέ μεταξύ ε, τη προανατολική και τη προανατολική Γερμανία, βλέπω να έχουμε στην ε, συνολική παραγωγικότητα της εργασίας στην δική μας Ανατολική Γερμανία ε, πολύ πιο δύσκολες συνθήκες και μάλιστα επιδείνωση των συνθήκων, επιδείνωση παραγωγικότητας. Άρα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την απασχόληση, να αμύψουμε σωστά τη δουλειά, όσο ωραίο και αν φαίνεται όμως αυτό, δεν έχουμε βρει τον τρόπο να το πράξουμε. Ερωτώ λοιπόν αν έχετε κάποιες λύσεις για όλα αυτά και για το πώς θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί η κοινή γεωργική πολιτική κατά τρόπον ώστε να απαλλαγεί και από το ε, γραφειοκρατικό άχθος που τη χαρακτηρίζει. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, ακούσαμε μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση και προτάσεις. Και έχουμε φυσικά και προτάσεις και υποδείξεις από πολλές πολιτικές ομάδες τα τελευταία χρόνια και από τη δική μας από ό,τι μας είπατε, αναλύσετε τις προτάσεις αυτές με τους συναδέλφους σας και η σύστηση αυτή κάνει ορισμένε συστάσεις στα κράτη-μέλη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στο μέλλον φαίνεται ότι θα υπάρξει υποστήριξη της παραγωγής παρόμοια σε όλα τα κράτη-μέλη η οποία σχεδόν ενιαία θα χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό της Ένωσης. συμμερίζουμε σε μεγάλο βαθμό την ιδέα αυτή, αλλά είπατε μια σημαντική φράση. Είπατε, αν δούμε τα, τις ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις, θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα ορισμένο ποσό για μια γεωρική εκμετάλλευση χωρίς να έχουμε έναν τόσο πολύπλοκο μηχανισμό υποστήριξης όπως αυτό που έχουμε τώρα ή στις παλιότερες κράτη-μέλη. Θα μπορούσατε να το αναπτύξετε λίγο το θέμα αυτό γιατί συνδέεται με κάτι άλλο. Με ένα άλλο ερώτημα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ενιαία πληρωμή και ενιαία εφαρμογή. Αίτηση που σημαίνει μείωση στην γενικότερη γραφειοκρατία η οποία βαρύνει τα κρατημέλη και την Ένωση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο αναφέρθηκε η λειτουργία της υπαίθρου. Θέλουμε η έπεθρος να έχει ανθρώπους, θέλουμε ανθρώπους να ζουν και να εργάζονται στην υπαίθρο και δεν χρειαζόμαστε μόνο άμεση ενίσχυση στην παραγωγή για τους γεωργούς. Χρειαζόμαστε επίσης και καλύτερη ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών. Καλά σχολεία, καλή ιατρική κάλυψη, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κατά κάποιο τρόπο αναφερθήκατε σε προγράμματα του δεύτερου πυλώνα που συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου και τα σχόλιά μου και οι ερωτήσεις μου. Και ξανατονίζω ότι το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μελλοντική δουλειά μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία Ροβάη. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα σχόλια του κύριου Μπλάτφερντ ότι στη Γεωργία τα δημόσια αγορά αγαθά παράγονται όταν παράγεται υπάρχονται τρόφιμα. Το να μιλάμε για το σε τι βαθμό η γεωργία συμβάλλει στα δημόσια αγαθά δεν έχει νόημα μόνο το σεβασμό που έχω στον ομιλητή δεν συμφωνώ με το σημείο αυτό. Όντως η παραγωγή τροφίμων έχει ορισμένες επιπτώσεις. Ορισμένα σε ένα βαθμό παράγουν δημόσια αγαθά, ορισμένα λιγότερα. Λιγότερα όταν έχουμε παραγωγή σε τεράστια κλίμακα όπου χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα, χρησιμοποιούνται μηχανήματα από πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι υπέρ του δημόσιου προϊόντος, είναι υπέρ της κερδοφορίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που παράγουν ορισμένα προϊόντα ενώ οι μικροί αγρότες και οι μεσαίου μεγέθους ε, αγρότες, οικογενειακά αγροτήματα, αυτοί όταν παράγουν τρόφιμα, το τρόφιμο αυτό είναι δημόσιο αγαθό. Μετά έχουμε μεταφορά του προϊόντος, καταστρέφοντας τη φύση στη διάρκεια της μεταφοράς, καταστρέφοντας το περιβάλλον πολλές φορές, αυτό δεν συμβάλλει στη δημιουργία δημόσιων αγαθών, παρότι παράγεται και πωλείται τροφή. Και πιο μεγάλη είναι η συμβολή στα δημόσια προϊόντα όταν η παραγωγή στηρίζεται στην τοπική παραγωγή, στις τοπικές πωλήσει, στην επιτόπια επεξεργασία του προϊόντος, νοπά προϊόντα, πολύ καλής ποιότητας, στην τόπια αγορά. Γι' αυτό όλα αυτά τα σχόλια θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλάμε για τη νέα βάση του συστήματος ενιαίων πληρωμών. Ευχαριστώ. Vă mulțumesc. Am să dau acum cuvântul domnului Biro pentru a răspunde întrebărilor adresate. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Biro για τις απαντήσεις του. Παρακαλώ. Merci. Ε, ευχαριστώ. Μου αναφέρατε τόσα πολλά θέματα που με δυσκολία μπορώ να, να τα ξαναβρω. Ένα σημείο που αναφέρατε πολύ και κατά τη γνώμη μου όχι και τόσο μπερδεμένο είναι το θέμα της ε, ΠΟΕ. Αρκετοί μιλήσατε για την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Μα οι συμφωνίες της ΠΟΕ δεν θα παίξουν ιδιαίτερα στο σύστημα αμέσων ε, ενισχύσεων, ακόμη και αν έχουμε συμφωνία στην ΤΟΑ. και η συμφωνία δεν θα είχε παρά στη μείωση των ε, τελών ε, και των δασμών ε, για, τα, για την κτηνοτροφία. Αυτό θα ήταν το πιο επικίνδυνο. Δηλαδή οι γαλακτοφόρες αγελάδες θα είναι αυτές που θα υποφέρουν περισσότερο από κάτι τέτοιο. Τώρα θα πρέπει να να πάρουμε τις ε, άμεσες ε, πληρωμές ε, και να τις συνενώσουμε στην περίπτωση των γαλακτοφόρων αγελάδων θα ήταν ενδιαφέρον. Βλέποντας δηλαδή και την εισοδηματική ενίσχυση και την περιφερειοποίηση και οι περιφέρειες που θα δουν ποια συστήματα είναι αυτά που πρέπει να ενισχυθούν ή στα πλαίσια ενός δεύτερου, του δεύτερου πυλώνα που μόλις ανέφερα για πιο περιφερειοποιημένα συστήματα. Εκεί μόνο μπορούν να χρησιμεύσουν οι πληρωμές, εκτός πια και αν μπουν μέσα στο πράσινο κουτί στην ΠΟΕ, οπότε θα έχουμε πρόβλημα με το περιθώριο χειρισμών που θα έχουμε. Δεν βλέπω λοιπόν μεγάλους κινδύνους να έρχονται από εκεί για το σύστημα των αμέσων ενισχύσεων στο βαθμό δηλαδή που το πράσινο κουτί δεν θα αφισβητηθεί και αν δεν γίνει και τη ρυθμική προσαρμογή των πληρωμών εκτός πια και είναι μικρά τα ποσά όπου θα έχουμε δηλαδή αντικυκλικές πληρωμές. Άλλοι αναφερθήκατε στη ζωντάνια της Υπέθρου, στην απασχόληση στην υπαίθρο και να έχουμε πληρωμές που θα λαμβάνουν υπόψη τους εργαζόμενους. Άλλοι είπατε ότι ανεκτάριο θα δημιουργούσε πρόβλημα <coughs> για τις εκτός εδάφους παραγωγές, γιατί δεν θα ήταν επιλέξιμες αυτό λοιπόν που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα μεταξύ κρατών μελών είτε για τις, ε, ε άμεσες, ε, για τις ενιαίες πληρωμές ε, στα πλαίσια των 27 ή των κρατών μελών. Και αν μιλήσουμε εμείς για ενισχύσεις εκτάριο υπάρχουν παραγωγές θερμοκηπίου που δεν θα ενισχυθούν ούτως ή άλλως δεν ενισχύονται ιδιαίτερα σήμερα Το κριτήριο λοιπόν πληρωμής ανά έκταρο μας φαίνεται το λιγότερο κακό διότι θα βοηθήσει πιο εντατικές παραγωγές και ξέρουμε ότι υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ εντατικής γεωργίας και ε, παροχής δημοσίων αγαθών. Βέβαια αυτό μόνο πολυμερικώς θα διορθώσει αυτές τις ανισότητες γιατί πιο πολλά εκτάρια έχετε πιο πολλά λεφτά παίρνετε. Οπότε Εμείς ε, χρησιμοποίησαμε έναν ε, συντελεστή, τον συντελεστή του Τσίνη για να μπορέσουμε να περάσουμε από, ε, να, μειώσουμε μάλλον τις εισοδηματικές ανισότητες. Αυτό είναι πιο προασπίσιμο από ότι εναλλακτικέ λύσεις τύπου της ιστορικής βάσης που χρησιμοποιούν ορισμένα κράτη ή ανακμετάλλευση. Σήμερα είναι τόσο ετερογενής η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τεράστιες γεωργικές επιχειρήσεις στη Γερμανία ή στη Σλοβακία, ενώ σε άλλα κράτη οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι πολύ μικρές. Θα πρέπει να γίνεται λοιπόν καταβολή αναμισθωτό, ανεργαζόμενο. Βέβαια εδώ έχουμε ένα παράδοξο αποτέλεσμα, δηλαδή αν εμείς τον τωρινό προϋπολογισμό διατηρώντας και περιφερειακούς ε, φακέλους ε, για να αποφύγουμε τις, ε, τα αποτελέσματα μεταφορών μεταξύ των περιφερειών, αν εμείς πληρώσουμε ανεργαζόμενο δεν μειώνουμε τις ανισότητες. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα πλαφόν ανεργαζόμενο και καταβολή ανεκτάριο. Βέβαια αυτή η οροφή είναι δύσκολο να καθοριστεί και αν ορισμένα κράτη το θέλουν σε επίπεδο εθνικής επικουρητότητας να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα, να βάλουν κατόφλια ε, για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, γιατί αν εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα δεν είναι κακό να έχουμε οροφές ανά άτομο. Αυτό βέβαια λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ανέφεραν την ανταγωνιστικότητα. Ένα ενιαίο σύστημα καταβολών ανεκτάριο δεν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα ανταγωνιστικότητας τουλάχιστον έναντι της τωρινής ΚΑΠ τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας μπορούν να προκύψουν είτε από τις δομές σε ορισμένες χώρες έχουμε πάρα πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις που δεν θα πρέπει ντε και καλά να τις διατηρήσουμε διότι θα έχουμε μικρές δυνατότητες παραγωγής και που δεν θα μπορούν να συντηρήσουν έστω και έναν μερικό απασχολούμενο εργαζόμενο. Σήμερα με την αποσύνδεση Έχουμε τεράστια γραφειοκρατία τουλάχιστον στη Γαλλία. Αλλά αυτοί που επιβάλλουν σήμερα την γραφειοκρατία είναι αυτοί οι οποίοι φωνασκούν περισσότερο κατά της γραφειοκρατίας και η Γαλλία είναι το ιδανικό παράδειγμα διότι εμείς επιλέγουμε τις πιο μπερδεμένες και πιο γραφειοκρατικές ε, λύσεις ε, για τη χώρα μας ε, πράγμα που δεν εμποδίζει την, κυβέρνηση να ασκεί κριτικές στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε προβλήματα για τους ε, Ευρωπαίους ε, γεωργούς ε, έναντι των άλλων χωρών και αυτό είναι το κόστος, το κόστος της εργασίας και όχι μόνο και στη Γεωργία αλλά και αλλού και έχουμε και κανόνες ότι η κοινωνία ζητάει συνεχώς πιο δεσμευτικές, έχει συνεχώς μάλλον πιο δεσμευτικές απαιτήσεις. Ας πούμε για τη ρουσμή γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ε, ε, ας πούμε το μη τροποποιημένο καλαμπόκι το αγοράζαμε κατά 30% πιο ακριβά από ό,τι από άλλες ε, χώρες που επιτρέπουν το καλαμπόκι, το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. Πρέπει λοιπόν εμείς να αντισταθμίσουμε αυτά τα μειονεκτήματα. Τώρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μιλήσατε για τη βιωσιμότητα ε, ε, της υπαίθρου ε, που δεν, και τα προβλήματα που θα προκύψουν αν δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι πτυχές. Ένας από τους μεγάλους κινδύνους άμα καταργηθεί η ΚΑΠ δεν είναι μόνο το θέμα της ανταγωνιστικότητας ούτε το ρίσκο ότι δεν θα έχει φαΐ ο πλανήτης ε, ε, ε, εάν υπάρχει μία πραγματική ζήτηση θα αυξηθούν οι τιμές και η παραγωγή θα ακολουθήσει. Ο πραγματικός κίνδυνος εξαφάνισης της ΚΑΠ και και των πληρωμών είναι να έχουμε εγκατάλειψη των γεωργικών περιοχών, να έχουμε συγκέντρωση γεωργικών περιοχών με αρνητικά αποτελέσματα και σε επίπεδο περιβάλλοντος αλλά και να διατηρήσουν αλλά και η διατήρηση του πληθυσμού της υπαίθρου στον τόπο τους είναι ένας στόχος. Εμείς εδώ δεν κάνουμε συστάσεις ε, για τα κράτη-μέλη, εμείς ε, δίνουμε προσανατολισμούς από τον απολογισμό του τωρινού συστήματος και προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας και αυτή την πλευρά, δηλαδή να έχουμε ε, πληθυσμό στην ε, Ήπεθρο, ε, να πληρώνεται η παρουσία αυτού του πληθυσμού για την παραγωγή δημοσίων αγαθών. Διάφοροι stakeholders συμμετείχαν σε μια ομάδα της Κομισιόν για την Ανάπτυξη της Υπέθρου. 12 σημεία έχουν ε, οριστεί από αυτήν την ομάδα στον ε, κατάλογο των ε, παροχών κοινή ωφελία των δημοσίων αγαθών που προσφέρει η περιβάλλον, νερό κλπ. Θα μπορούσαμε εμείς να εργαστούμε πάνω σε αυτόν τον κατάλογο αλλά αυτές τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια θα πρέπει να τις χρηματοδοτήσουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανές, να εγγυθούμε βιωσιμότητα ε, στην Ήπεθρο. Τώρα, για να ενώσουμε το, τους πυλώνες 1-2 εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν προβληματισμό σχετικά με τη γενική δομή της ΠΑΚ. Αν ε, σήμερα λάβουμε υπόψη όλη αυτή την ευελιξία που ανέφερα άρθρο 68 για την ενίσχυση των ευπαθών παραγωγών κλπ. Ε, κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και στο δεύτερο πυλώνα. Το όριο μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα, αν το κοιτάξουμε καλά, είναι δύο ε, ε, στυλ. Αφενός έχουμε την διοικητική ε, διαφορά μεταξύ των δύο πυλώνων όπου θα έπρεπε λόγω απλούστευσης να έχουμε μια ενιοποίηση της διοικητικής διαδικασίας και μετά μέτρα τα οποία έχουμε στο δεύτερο πυλώνα και τα οποία ε, μπορούν να πλουστευτούν πηγαίνοντας στον πρώτο πυλώνα και που ήδη δηλαδή πάνε στον πρώτο πυλώνα χρησιμοποιώντας το άρθρο 68 όπως κάνει η Γαλλία. Για το σενάριο τώρα συγχρηματοδότησης η διάκριση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα είναι μια καθαρά διοικητική διάκριση και δεν αποκλείεται να περάσουν ε, ε, βρείτε τα ε, προγράμματα για την πληρωμές στις μειονεκτικές περιοχές αν θεωρήσουμε ότι δεν χρειάζεται η α ή β δημοσιονομ... ο α ή ο β δημοσιονομικός προγραμματισμός. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται πολύ μπερδεμένα, αλλά από εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να σκεφτούμε εμεί ε, μία δομή πολύ πιο συνολική, χωρίς ε, ε, να αναρωτιόμαστε τι θα μπαίνει στον πρώτο ή στον δεύτερο πυλώνα. Κάτι άλλο το οποίο ετέθη είναι το θέμα της χρηματοδότησης από τον πρώτο πυλώνα. Είναι κάτι το προβληματικό, υπήρχε μεγάλη ασυμφωνία στην ομάδα των πανεπιστημιακών που συνέταξαν αυτή την έκθεση ασυμφωνία που νομίζω ότι ε, βασιζόταν και στην εθνικότητα των μελών αυτής της Επιτροπής. Είναι δύσκολο και σε θεσμικό επίπεδο αν είχαμε έναν συγχρηματοδοτούμενο πρώτο πυλώνα, δεν μπορούμε εμείς ε, να υποχρεώσουμε ε, κοινοτικές δαπάνες σε ένα κράτη-μέλη, διότι σημαίνει ότι τα υποχρεώνουμε σε δαπάνες ε, στον εθνικό προϋπολογισμό, δηλαδή παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία. Θα έπρεπε να έχουμε ένα συνολικό προϋπολογισμό και ένα εθνικό φάκελο ιδέες ρίχνουμε, δεν λέω ότι έχουμε τη λύση. Αλλά σε αυτόν τον φάκελο θα μπορούσαν να προσφεύγουν τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση του α του β μέτρου. Υπάρχει όμως ένας ε, κίνδυνος ε, να έχουμε μια πολιτική που θα είναι ένα και λιγότερο κοινή. Και μερικοί ρώτησαν με σε τέτοια περίπτωση θα παραμείνει κοινή η ΚΑΠ. Εγώ λέω ότι χρειάζεται να έχουμε κοινούς ε, κανόνες για το τι εστί κοινή ωφέλεια, για το τι ένα κράτος μπορεί να κάνει, αλλά σήμερα έχουμε μία κατάσταση όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο και εδώ μιλάω εκφράζοντας την προσωπική μου γνώμη και όχι της ομάδας, να φανταστούμε μία γεωργική πολιτική ε, λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των δομών, των γνωμών, ε, του βιωτικού επίπεδου των γεωργών με στα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολο λοιπόν να κάνουμε κάτι που να μην βασίζεται ιδιαίτερα σε μια ενισχυμένη αρχή της επικουρικότητας. Χρειάζονται λοιπόν κανόνες όπου να μην έχουμε περιπτώσεις χρηματοδότησης μια συγκεκριμένης δράσης σε μια χώρα που σε άλλη δεν χρηματοδοτείται. Πρέπει λοιπόν να ε, έχουμε ένα απόλυτα κοινό πλαίσιο από νομοθετικής πλευράς. Δεν είμαι σίγουρος ε, για το κατά πόσο ξέχασα ή όχι. Με δυσκολία παρακολούθησα πολλούς από τους ερωτούντες. Δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάτι. Αν έχετε να με ρωτήσετε, είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ευχαριστώ κύριε Μπιωγό για την παρουσίαση αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας έκθεσης και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Νομίζω ότι το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων είναι κάτι το οποίο θα επανεξετάσουμε και σε άλλες μας συζητήσεις και χρειάζεται μεγάλη συνένεση σχετικά με αυτό το καθεστώς για να μπορέσουμε η μελλοντική ΚΑΠ να έχει μια νομιμότητα που εμείς ε, θέλουμε και να αναγνωριστεί και από το κοινό. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα ψηφίσουμε την έκθεση για τη γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, ειδικό έλεγχο της ε, υγιούς λειτουργίας. Έχουμε 80 τροπολογίες, εισηγητής είναι ο κύριος Ντόρφμαν. Και ο κύριος Ντόρφμαν προτείνει μερικούς συμβιβασμούς. Ε, είστε έτοιμος κύριε Ντόρφμαν να μιλήσετε. Ähm, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εδώ έχουμε μια έκθεση να ψηφίσουμε, την οποία έχουμε ήδη συζητήσει δύο φορές στην Επιτροπή μας. Ως προς το περιεχόμενο είναι όχι εύκολη η υπόθεση αυτή. Έχουμε τεχνικά ζητήματα που πρέπει να προσδιορίσουμε για τα κριτήρια των ε, περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα. Και ναι μεν γνωρίζουμε το, τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει στήσει και τις προσωμιώσει από τα κράτη-μέλη, Προσωμιώσει που θα έπρεπε να έχουμε λάβει, αλλά δεν τις έχουμε δει ακόμη. Δεν έχουμε γνώση των προσωμιώσεων αυτών και ω εκ τούτου θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να αποφύγουμε κρίση ως προς το, ε, τα ποσοτικά στοιχεία των κριτηρίων, κυρίως τα τις οριακές τους τιμές. γιατί έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή να μας δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι λοιπόν και από όσο εγώ γνωρίζω, τέτοια κριτήρια σαν αυτά που θέλει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγούν σε τέτοιες ε, πιές, αυτές τις, ε, πιο, τις ε, μειονεκτούσες περιοχές, τις περιοχές με τα φυσικά μειονεκτήματα που δεν θα τους επιτρέψουν να ε, λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία και για τις συζητήσεις και τις προσπάθειες να προαγάγουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες έτσι ώστε η έκθεση αυτή να εγκριθεί από το σώμα και να είναι μια καλή έκθεση εν τέλει. Ευχαριστώ. Λέω ο Πρόεδρος, περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Υπάρχει μόνο ανατροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες Εγκρίνεται. Υπαριθμών 2. Τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίες Εγκρίνεται.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 Βρείτε μια άλλη θέση αν δεν δουλεύετε με χάρη με αυτό. peut continuer Amendement 3. Υπαριθμόν 3. Τροπολογία. Άρχεται ψηφοφορία. Παρακαλώ. Le vote est clos. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Υπαριθμών 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Υπάρχει μία ψήφος παραπάνω από το ΕΛΚ. Να επαναληφθεί η ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την υπαριθμόν 12 τροπολογία. σου. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 11, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε Απορρίπτεται. 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Υπάρχει μόνο 20, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα στις σωφορίες. Thank you. Υπαριθμόν 22, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 23. τρία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Η 29 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 30 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 31 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της προφορίας εγκρίνεται. 38 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 41 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της προφορίας απορρίπτεται. 39 άρχεται η ψηφοφορία. Κλο. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 40 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Η 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρες της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 45 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 46 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 47 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της προφορίας εγκρίνεται. 48 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφορίας εγκρίνεται. Η 50 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφορίας απορρίπτεται. Η 52 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 49 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 51 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54. Όχι. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. 55. πέρασε τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 3 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 65. Όχι. 63 λέει ο πρόεδρος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 65. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 66 Πέρας. Απορρίπτεται. 67, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 70, άρχεται η ψηφοφορία. 70. Πέρας. Απορρίπτεται. 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 73 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 74 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Υπαριθμόν 4 συμβαστική παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική παριθμών 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 86. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 88 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 89 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 90 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Στην 92 του κυρίου Σμιτ υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ κύριε Σμιτ πείτε μας τι θέλετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε φτάσει στο τέλο αυτή τη ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να προσθέσουμε στο κείμενο απαιτεί την προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Δεδομένων και των επερχομένων συζητήσεων για τον προπολογισμό, που θα χρειαστεί να υπάρχουν και αυτές, αυτοί οι προσδιορισμοί, γιατί και θα δούμε και τι τεχνικέ λεπτομέρειε. Ελπίζουμε να μα υποστηρίξουν οι συνάδελφοι. Ο Πρόεδρο, έχει κανεί αντίρρηση ω προ την υποβολή σε ψηφοφορία αυτή τη προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 92, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Και εγκρίνεται. Και τώρα σας παρακαλώ να ψηφίσουμε τις συστάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής. Πρώτο, Γνωμοδότηση, μάλλον, εννοεί ο Πρόεδρος. πέρα τη ψηφοφορία Απορρίπτεται. υπαριθμόν 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. υπαριθμόν 10 στη γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ε, σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Από το ΕΛΚ έχουμε μία ψήφο παραπάνω. Ας επαναλάβουμε την ψηφοφορία λοιπόν. Επαναλαμβάνουμε την πρόταση του τροποποιημένου κειμένου. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Καμία ψήφος κατά. Δύο αποχές. Συγχαρητήρια στον Σίγητη. Και περνάμε. Nous allons procéder au vote σε ψηφοφορία της έκθεσης πρωτοβουλίας για την απλοποιημένη ΚΑΠ. Εισηγητής Άσουαρθ. 230 τροπολογίες. Επαναλαμβάνω εισηγητής ο κ. Ρίτσαρντ Άσχορθ, 230 τροπολογίες. Ο ζητητής θέλει να κάνει εισαγωγή. Η κυρία Εράνση. Ε, ήθελα να πω ότι στην τροπολογία 188 ο συνάδελφος Μάτο και εγώ βγάζουμε τις παραγράφους ε και F, ε σίγμα τάφ στα ελληνικά, από τις τροπολογίες του ΕΛΚ. Βγάζουμε λοιπόν το ε ή το F και το F ή αν θέλετε αλλιώ το 3 ή 4. On passe euh, au vote. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Ξέχασα να σας πω, ξέχασα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, αν θέλει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι στην έκθεση αυτή αυτό που σκόπιμα θέλουμε να κάνουμε είναι να ορίσουμε αρχές που θα περάσουν στην ε, μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ, αρχές για απλοποίηση της ΚΑΠ, αρχές για να είναι πιο εύκολη η ζωή των γεωργών. Το λέω αυτό διότι μερικές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, ουσιαστικές τροπολογίες που ανήκουν την έκθεση μεταρρύθμισης της ΚΑΠ του Τζον Λάινον όχι στην έκθεση για την απλούστευση. Είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό σε μερικά σημεία λέω όχι σε αυτές τις τροπολογίες. Όχι γιατί συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά διότι θέλω να τονίσω ότι οι τροπολογιστές δεν ανήκουν σε αυτή εδώ την έκθεση. Ανήκουν στην έκθεση στην ψηφοφορία για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠΑ. Πρόεδρος, ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 1. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Συγγνώμη, τροπολογία 2. Ψηφίζουμε, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ψηφί, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 1. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκατρία. Έναρξη. Και λήξη. Απορρίπτεται. 14 έναρξη και λήξη εγκρίνεται 15 έναρξη λήξη εγκρίνεται 16 έναρξη Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 2. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 25. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 26 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται 27 έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 28 έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 29. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 30. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 31. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 32. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 33. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 34. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 35 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 36. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 37. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική παραθμόν 3. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Σαράντα οχτώ. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Σαράντα εννέα. Έναρξη. Λήξη. Απορρίφθηκε. 50 έναρξη λήξη απορρίβεται 51 έναρξη όχι 52 51 51 έναρξη λήξη απορρίβεται 52 έναρξη λήξη εγκρίνεται 53 έναρξη λήξη απορρίπτεται 54 έναρξη λήξη εγκρίνεται 56. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 57. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 58. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 75. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 76. Ε, έναρξη. λήξη απορρίπτεται 77 σε δύο τμήματα πρώτο έναρξη λήξη εγκρίνεται δεύτερο τμήμα έναρξη λήξη απορρίπτεται 78 έναρξη λήξη εγκρίνεται 79 έναρξη λήξη εγκρίνεται 80 έναρξη λήξη απορρίπτεται 81 έναρξη Λήξη. Εγκρίνεται. 82. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 83. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 84. Έναρξη. λήξη απορρίπτεται 85 έναρξη λήξη απορρίπτεται 86 έναρξη λήξη εγκρίνεται 87 έναρξη λήξη εγκρίνεται 88 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα έναρξη λήξη εγκρίνεται και δεύτερο τμήμα έναρξη λήξη απορρίπτεται 89 έναρξη λήξη απορρίπτεται 90 έναρξη λήξη εγκρίνεται 91 έναρξη λήξη εγκρίνεται 92 έναρξη Λήξη. Εγκρίνεται. 95. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 96. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 97 έναρξη κλίξη εγκρίνεται 100 έναρξη κλίξη εγκρίνεται 102 έναρξη λήξη εγκρίνεται 103 έναρξη λήξη απορρίπτεται 105 έναρξη λήξη εγκρίνεται 107 έναρξη λήξη εγκρίνεται 108 έναρξη λήξη απορρίβεται 109 έναρξη λήξη εγκρίνεται 110 έναρξη λήξη εγκρίνεται 111 έναρξη λήξη απορρίπτεται 112 έναρξη Λήξη. εγκρίνεται. Συμβαστική προθυμών 4. Έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται. 118. Έναρξη. Λήξη εγκρίνεται. 119 έναρξη λήξη εγκρίνεται 120 έναρξη λήξη μία ψήφος επιπλέον σοσιαλιστών. Ξαναψηφίζουμε την 120. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. 121. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 122. Έναρξη. 126. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται η 126. 127. Έναρξη. λήξη απορρίπτεται 128 έναρξη λήξη εγκρίνεται 129 έναρξη λήξη εγκρίνεται 130 έναρξη λήξη εγκρίνεται 131 έναρξη λήξη εγκρίνεται 132 έναρξη λήξη εγκρίνεται 133 έναρξη λήξη απορρίπτεται 134 έναρξη λήξη απορρίπτεται 135 έναρξη λήξη εγκρίνεται 136 έναρξη λήξη απορρίπτεται 137 έναρξη λήξη εγκρίνεται 139 έναρξη λήξη εγκρίνεται 141 έναρξη λήξη εγκρίνεται 142 έναρξη λήξη εγκρίνεται 146 έναρξη Λήξη. Εγκρίνεται. 148. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 149. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Έναρξη. λήξη εγκρίνεται 165 έναρξη λήξη εγκρίνεται 166 έναρξη λήξη εγκρίνεται 167 έναρξη λήξη απορρίπτεται 168 έναρξη λήξη εγκρίνεται 169 έναρξη λήξη εγκρίνεται 170 έναρξη λήξη εγκρίνεται 171 έναρξη λήξη απορρίπτεται 172 έναρξη

Λήξη. Εγκρίνεται. 179. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 180. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 181 έναρξη λήξη εγκρίνεται 182 έναρξη λήξη εγκρίνεται 183 έναρξη Λήξη εγκρίνεται. 185. Έναρξη. Τεχνικό πρόβλημα. θα πρέπει να ψηφίσουμε τα χέρια γιατί κάποιο μηχάνημα δεν λειτουργεί. Ψηφίζουμε την 185 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 186 υπέρ. κατά εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ. Κατά. εγκρίνεται 188 πρώτο τμήμα υπέρ κατά Φαίνεται ότι αλλάξετε γνώμη στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ξαναρωτάω. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. 2020. Εγώ δεν ψήφισα, άρα εγκρίνεται. Τα ψηφίσω κι εγώ, είμαστε 21. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Πέμπτο τμήμα της τροπολογίας 188. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. 21 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. κατά εγκρίνεται Συμβαστική 7 υπέρ Καταρχήν ο κύριος Γκλάτφελντ ζήτησε το λόγο. σχετικά με την ε, συμβαστική υπαριθμών 7. Είναι συμβατή με την 111 που ανεφέρεται σε εγωπρόβετα ε, νεότερα των 12 μηνών. Να μην πάνε στο προσφαγείο. για εγωπρόβατα κάτω από την ηλικία των 12 μηνών. Να μην εντοπίζονται ηλεκτρονικά, να μην υπάρχει ηλεκτρονική σήμανση. Nous Ελπίζουμε τη συμβαστική υπαριθμών 7 υπέρ κατά 215 υπέρ. Qui est contre Κατά. Απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται.

Εγκρίνεται. 220 υπέρ. Qui est contre Κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. συγκρίνεται. 222 υπέρ κατά εγκρίνεται 223 υπέρ κατά εγκρίνεται 228 υπέρ κατά εγκρίνεται 229 υπέρ κατά εγκρίνεται 230 υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ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 Συγχαρητήρια στην εισηγητή. Με 29 υπέρ, κανείς κατά 10 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Άσκορφ.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 το επόμενο σημείο αφορά στο δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας ανεφοδιασμού για την Ευρώπη. Ο Ζωζέ Μποβέ έκανε αυτή την έκθεση. Ο κύριος Πιέρ Λουίτζι Λοντέρο εκπροσωπεί την Κομισιόν και δίνω το λόγο τώρα στον Ζωζέ Μποβέ, ο οποίος εξετάζει το θέμα της τιμής των τροφίμων. Καλημέρα σε όλους. Εμείς ε, θα συζητήσουμε για πρώτη φορά το έγγραφο εργασίας που αφορά στο δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και μια λυσίδα, ε, πιο αποτελεσματική αλυσίδα ανεφοδιασμού στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε, αυτήν, όλη αυτή τη συζήτηση με ένα έγγραφο εργασίες, ούτως ώστε ο καθένας από εσά, αφού το διαβάσει να μπορέσει να κάνει ερωτήσεις, να μιλήσει, να κάνει παρατηρήσεις και μετά να συντάξουμε αυτή την έκθεση, να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και στη συνέχεια να καταφέρουμε, ελπίζω, να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση. Η θέμα, το, θέμα ετέθη λόγω μιας εργασίας που έκανε η Κομισιόν και που μας ε, ε, ε, υποδεικνύει ορισμένα προβλήματα προβλήματα τιμών, προβλήματα τροφιμικής αλυσίδας, διαφάνειας για τις τιμές, σχέση μεταξύ υπεραξίας όπως κατανέμεται στην από την παραγωγή στη μεταποίηση και πώς φτάνει στην διανομή. Κάνει αναφορές σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αγρότης από το 31% που έπαιρνε το 95% παίρνει 26% το 2005 και άμα το κάνουμε και μια προβολή στο 2010 ακόμη πιο χαμηλά θα είναι τα ποσοστά του Γιωργού. Αυτό λοιπόν θέτει και όλη την προβληματική για το γεωργικό εισόδημα. Έχει να κάνει με την αναδιοργάνωση της ε, γεωργίας, ε, με την οργάνωση τροφιμικής αλυσίδας, ε, με την πολιτική των σούπερ μάρκετ κλπ. Δεν θα σας τα ξαναδιαβάσω όμως από το κείμενο, θα σας πω άλλα πράγματα. Σήμερα έχουμε, μια μεγά, έχουμε μεγάλες διαφορές στη Γεωργία. Έχουμε 14.600.000 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη που απασχολούν 12.500.000 άτομα. Έχουμε πάρα πολλούς λοιπόν γεωργούς αλλά με τεράστιες διαφορές στην υποστήριξη που τους δίνεται. Και αυτό γιατί μόνο το 0,02% των εκμεταλλεύσεων παίρνουν πάνω από 300.000 ευρώ ενίσχυση, ενώ το 77% παίρνει κάτω από 5.000 ευρώ. Βλέπετε τις ανισότητες λοιπόν και τις επιπτώσεις φυσικά που έχουν. Σε επίπεδο επιχειρήσεων έχουμε ε, μεταποιητικές ε, επιχειρήσεις με μεγάλες ανισότητες επίσης. Έχουμε μεγάλες ε, βιομηχανίες, εθνικές είτε υπερεθνικές και απ' την άλλη έχουμε πάνω από 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μικρές οι οποίες βρίσκονται στον τομέα των τροφίμων. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη συγκέντρωση από τη μια και από την άλλη ένα σωρό μικρά εργαστήρια μεταποίησης και οι σχέσεις μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή δεν είναι πάντα ίδιες. Η Νεστλέ έχει ένα τζίρο 70 δις ευρώ, η Ντανόν 15 2 είναι οι δύο πιο, πιο μεγάλοι, 11,2 δις ε, κέρδη ε, για την Εστλέ ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ε, μία απόδοση 1 με 2% ε, το χρόνο κατανομή εισοδήματος σε μετόχους ή ιδιοκτήτες ενώ η Νεστλέ μοιράζει μερίσματα της τάξης του 14% και εντανών του 11,8%. Βλέπετε λοιπόν την τεράστια διαφορά. Δηλαδή επίσης στον τομέα της διανομής και εδώ η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σύνθετη έχουμε από τη μια τα μικρά μπακάλικα τα οποία σήμερα είναι θύματα ε, τις, ε, και τίνουν προς εξαφάνιση και από την άλλη έχουμε μία μεγάλη συγκέντρωση. Βλέπουμε ότι οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, της διανομής έχουν και το 66% των πωλήσεων στα χέρια τους στην Ευρώπη. Δηλαδή άμα πάρουμε πάλι τα νούμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάρουμε τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ορισμένες χώρες, έχουμε πάλι συγκέντρωση. Έχουμε λοιπόν μία συγκέντρωση στη διανομή ε, των, ε, της ε, γεωργικής παραγωγής, 81% για τη Σουηδία, 80% για τη Γερμανία, 70, 80% ε, για τη Δανία, 70% για τη Δανία για την Γαλλία και την Γερμανία και 35% για την Ιταλία. Είδατε λοιπόν εσείς τις διαφορές μεταξύ λοιπόν παραγωγών μεταποίησης και διανομής. Υπάρχει το θέμα των ε, νόμιμων πρακτικών, δηλαδή ε, τι κάνουν αυτοί οι παραγωγοί όταν έχουν μπροστά τους την μεταποίηση και όταν έχουν απέναντί τους τη διανομή. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να σταθώ ε, σε όλες αυτές τις σχέσεις αλλά το πρόβλημα τίθεται σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων αυτών. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο το δακτυλοδεικνύει η Κομισιόν αλλά δεν έχει απάντηση. Είναι το θέμα της ε, πώληση με απώλεια ε, πώληση με ζημιά. Διότι ε, υπάρχει πρόβλημα, ανησυχούμε ιδιαίτερα, δεν υπάρχουν σήμερα νόμοι που είναι επιβεβλημένοι στις διάφορες χώρες και που να έχουν να κάνουν μεταξύ των λιανοπολιτών και του τελικού καταναλωτή. Σήμερα λοιπόν μπαίνει ένα κεντρικό ζήτημα. Δεν είμαστε εμείς ικανοί να ορίσουμε ποια είναι ε, η πώληση με ζημιά γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι η βασική τιμή ε, του γεωργικού προϊόντος ε, στην Ευρώπη και δεν μπορούμε λοιπόν να απαντήσουμε. Το θέμα λοιπόν της πώληση με ζημιά συνδέεται και μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή αλλά και μεταξύ αγρότη μεταποιητή, μεταποιητή και και σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και κάτι άλλο για το εισόδημα, ε, είναι η αυτοκατανάλωση. Η αυτοκατανάλωση είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην γεωργική παραγωγή. Δηλαδή, μία γεωργική παραγωγή που δεν περνάει μέσα από τα κανάλια της εμπορευματοποίησης. Και εδώ έχουμε στατιστικές για ορισμένες περιφέρειες. Η Ρουμανία είναι η χώρα η οποία έχει προχωρήσει και πιο μακριά για, στις στατιστικές για αυτό το θέμα, διότι 22% της τροφιμικής κατανάλωσης είναι αυτοκατανάλωση και δεν μπαίνει στο παραδοσιακό <coughs> κύκλωμα κατανάλωσης. Μας δίνει λοιπόν νέα στοιχεία αφορά σε μια σημαντική χώρα 23 εκατομμυρίων κατοίκων. Στις άλλες ε, χώρες ε, υπάρχουν τέτοιες πρακτικές με τους εργατικούς κήπους των πόλεων για παράδειγμα. Η Ήρα, το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωπονικής Έρευνας ε, στην Γαλλία, αποδεικνύει ότι το 22% της ντομάτας που καταναλώνεται στη Γαλλία είναι αυτοκατανάλωση οι ίδιοι καταναλωτές δηλαδή στους μπαξέδες ε, ε, στους οικογενειακούς τους μπαξέδες καλλιεργούν τις νομάτες. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με, τις, ε, με, τα κέντρα σύντησης ε, εκτός ε, οικογενειακής εστίας. Τι γίνεται τα συλλογικά συντηστικά κέντρα αυξάνουν το μερίδιό τους. Αν πάρουμε εμεί τις 15 χώρες της Ένωσης πριν από τη διεύρυνση, η πώληση κρέατος στις 15 χώρες είναι 25% της αγοράς. Ε, του παραγόμενου και εμπορευματευομένου κρέατος. Το 25% λοιπόν περνάει από την παραγωγή και την μεταποίηση στην ε, συλλογική σύντηση. Και αυτό πρέπει να μας αφορά όλους. Γιατί και εδώ στο κοινοβούλιο δηλαδή οι μεγάλες φίρμες, να αυτοί που μας ταΐζουν εδώ, στις Βρυξέλλες, ε, σερβίρει ένα εκατομμύριο τετρακόσες χιλιάδες γεύματα, δηλαδή 6 δισεκατομμύρια γεύματα το χρόνο στη Γαλλία. Δηλαδή φανταστείτε εσείς ε, το κομμάτι της αγοράς που έχουν στα χέρια τους. Και αυτή η επιρροή στην αγορά επηρεάζει και την αγορά και τις τιμές. Ένα άλλο στοιχείο που δεν λαμβάνεται υπόψη όταν φτιάχνουμε τις τιμές και που έχει να κάνει και με την πεταποίηση και την κατανάλωση είναι η απώλεια τροφίμων μέσα στην όλη αλυσίδα. Και έχουμε 240 κιλά τρόφιμα τα οποία πάνε στα σκουπίδια. Δηλαδή ο κάθε ε, αναευρωπαίο κάτοικο ε, πετάμε 240 κιλά τρόφιμα στα σκουπίδια, 200 ευρώ ανακεφαλή. Αυτά είναι νέα στοιχεία τα οποία τα χρησιμοποιώ για να σας δείξω πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα. Λοιπόν, τελευταίο στο τέλος του εγγράφου. Σας αναφέρω μερικά στοιχεία που θα επιτρέψουν να ανοίξουν τη συζήτηση και θα βοηθήσουν το Κοινοβούλιο να επεξεργαστεί προτάσεις και σε διαβούλευση με την Κομισιόν να προχωρήσουμε για να Είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Λοιπόν, η αοριστία των τιμών, το, το πάνω κάτω, το ανέβασμα-κατέβασμα των τιμών, διάρθρωση της τιμής, αλλά και διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία συνδέονται με υπερπαραγωγή που οδηγεί σε διαρθρωτικές μειώσεις Το είδαμε και με τη γαλακτοκομική κρίση. Η κερδοσκοπία για, την πρώτη, για τις πρώτες ύλες δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το θέμα, είναι διεθνές πρόβλημα. Όταν είχαμε πριν από 1,5 χρόνο την τροφιμική ε, κρίση οι τράπεζες τηλεφωνούσαν στους ιδιώτες ε, λέγοντας τους είστε έτοιμοι να επενδύσετε σε κερδοσκοπικά κεφάλαια πρώτων υλών. Ας πούμε σκέφτομαι εγώ το Credit Agricole, την ε, Γαλλική Αγροτική Τράπεζα που τηλεφωνούσε στους καταναλωτές κατευθείαν για να επενδύσουν σε κερδοσκοπικούς λογαριασμούς. Άλλο θέμα είναι ο ανεφοδιασμός, είναι σαφές το τι κάνουμε, δηλαδή να έχουμε καλύτερη ποιότητα και να είναι ευθέως ανάλογο με το εισόδημα των αγροτών. Είναι ένα θέμα που τίθεται πολλές φορές εδώ και για το κλίμα και για την ευημερία των ζώων, για τα θέματα που συνδέονται με το πετρέλαιο είναι θέματα πολύ σημαντικά. Τέταρτο είναι οι αηφόρες πρακτικές, οι δημόσιο, δημόσιος ανεφοδιασμός, αυτό σας τα είπα. Ε, άλλο θέμα που δεν συνδέεται άμεσα με το εισόδημα αλλά είναι σημαντικό για μας είναι πως μέσα από την επεξεργασία νέων γεωργικών πρακτικών που δεν μας επιτρέπουν να έχουμε υπερβολικό κόστος παραγωγής αλλά να είναι συμβατό με το σεβασμό της υπαίθρου, πώς αυτή η συζήτηση δεν προκαλεί την επιστήμη, τα ερευνητικά κέντρα, ούτω ώστε να εργάζονται πιο συμβατά, να συνεργάζονται με τους γεωργούς, να έχουν δηλαδή γεωργικά σχέδια τα οποία να είναι να εξοικονομούν ενέργεια, να σέβονται το περιβάλλον και να συνδέονται με όλες τις προβληματικές που έχουν να κάνουν με τη γεωργία και προστατεύουν το κλίμα. Είναι πολύ ανοιχτή η συζήτηση. Σήμερα δεν θέλω να φτάσω κατευθείαν με, με, προτάσεις. Εγώ θέλω να ξεκινήσει η συζήτηση, ο καθένας να εκφραστεί και μετά συλλογικά να επεξεργαστούμε και προτάσεις στα διάφορα κεφάλαια για τα οποία εμείς μπορούμε να παρέμβουμε στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ζωζέ, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ναι, για το έγγραφο αυτό. Οχτώ συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Κύριε Γκαρσία. Τι το πήρε στο... la ε, verdad es que es cierto lo que ha dicho el señor. Λοιπόν, η Κομισιόν μας παρουσιάζει για το ένα έγγραφο που αφορά στο... σε πολλά θέματα του παρελθόντος, ανησυχίες ε, που των παραγωγών και των καταναλωτών που είχαν δίκιο και που αποδείχτηκε δηλαδή ότι είχαν δίκιο με το έγγραφο της Κομισιόν και δόξα το Θεό δηλαδή διότι όταν ερχόντουσαν εδώ και καταγγέλανε όλη την ε, άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόταν νομίζαμε ότι λέγαν φαντασίες. Εγώ θεωρώ ότι η παρουσίαση του εισηγητή έχει μερικά κενά ε, έναντι του εγγράφου της Κομισιόν, δηλαδή το πώς θα ενισχύσουμε τα μέσα διαχείρισης της αγοράς. Αυτό μας οδηγεί σήμερα σε μια αστάθεια έντονη των τιμών και αυτό είναι γεγονός, όπως επίσης ε, και μειώνεται η διαπραγματευτική δυνατότητα των γεωργών μέσα στην όλη αλυσίδα. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν αυτά τα μέσα Επίσης ε, θα ήθελα να τελειώνουμε με την ανισορροπία μέσα σε αυτήν την αλυσίδα όπως και η Κομισιόν το θέλει. Αλλά για να κάνουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να είμαστε λογικοί και να μην δημιουργούμε συστήματα εθνικής ετικετοποίησης οι οποίες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, η γεωργική προσφορά μέσα από, συνεργασίες, μέσα από συνεταιρισμούς των γεωργών. Αυτές οι συμφωνίες οδηγούν στη διαχείριση της αγοράς και οδηγούν και σε σταθερότητα των τιμών. Θα πρέπει να διορθώσουμε την ε, νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και η ενιαία ε, οργάνωση, η κοινή οργάνωση των αγορών θα πρέπει να δίνει νομική υπόσταση σε, αυτές, σε αυτά τα συμβόλαια δια ε, επαγγελματικών οργανώσεων και οργανώσεων παραγωγών. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ε, είναι τα μικρά κυκλώματα εμπορευματοποίησης. Αυτό δίνει δυνατότητα να μειώνονται οι μεσάζοντες και δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα διαπραγμάτευσης στο γεωργό και μειώνονται και οι μεσάζοντες από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Επίσης, παρατηρητήριο τιμών θα αποτελούσε ε, θα, θα αποτελούσε έναν κορμό, ένα κλειδί όταν θα πρέπει να αναλύσουμε τις τιμές και να δούμε ποιες είναι οι ανισορροπίες στην τροφιμική λυσίδα. Και για να καταργήσουμε τις παράνομες πρακτικές που είναι κακές ε, και ζημιογόνες πρέπει να βρούμε και έναν μηχανισμό καταστολής για να σταματήσουμε την πώληση με ζημιά ε, ή την υπερτιμολόγηση. Επίσης ε, να έχουμε ε, κυρώσεις σε περίπτωση που δεν πληρώνουν ε, τα τιμολόγια αλλά και επίσης να μειωθούν οι προθεσμίες πληρωμής. Επίσης να εγγυθούμε τη σωστή πληροφόρηση του καταναλωτή ο οποίος δεν είναι πληροφορημένος πάντα σωστά και ένας κώδικας καλής πρακτικής για όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του ΕΛΚ, το λέω ως εισηγήτρια και συντονίστρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Λυπούμε που δεν θα μείνω στο τέλος της συζήτησης, αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητάνε ένα θέμα για το οποίο επίσης είμαι και ο Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος έχει λόγο. Κυρία, θα ήθελα να ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για την εκπόνηση αυτού του εγγράφου εργασία, το οποίο αποτελεί μια καλή βάση για την ε, διατύπωση ιδεών και ενό καλού μέσου για την εξασφάλιση το, της αλυσίδας, τη αλυσίδας ε, της ασφάλειας τροφίμων. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ε, έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουν και οι γεωργοί τις ε, θέσεις τους ε, για ένα εισόδημα ικανοποιητικό, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να είναι βιώσιμη η δουλειά τους. Ταυτόχρονα πρέπει και οι καταναλωτές να μπορέσουν να τοποθετηθούν. Πρέπει η δουλειά, τους, η δουλειά των γεωργών να βρίσκει την δίκαιη ανταπόδοσή της. θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για διαπραγμάτευση δηλαδή από αυτές τις ομάδες που καταπιέζονται, συμπιέζονται από την συντριπτική ισχύ των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν δηλαδή ε, τη δυνατότητα να προβάλλουν τα δικά τους επιχειρηματά τους. Και πολλές φορές είναι πολύ ψηλό το κόστος ή η επιπλέον επιβάρυνση για την ε, ε, διάθεση των προϊόντων τους και Επίσης θα πρέπει ε, να δούμε ποια σημεία, ποια κριτήρια θα είναι τα πιο σημαντικά. Η ποιότητα και η σχέση ποιότητας και τιμής ιδιαίτερα είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στα ανώτατα και τα κατώτατα επίπεδα, τις ε, οριακές τιμές δηλαδή. Γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε τις κερδοσκοπικές τάσεις. Δεν μπορούμε βέβαια να ε, αποτρέψουμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τη ελεύθερη διαμορφώση των τιμών. Ε, ωστόσο, ε, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι σπάνια η περίπτωση οι μεγάλε αλυσίδε των σούπερ μάρκετ να προμηθεύονται κατευθείαν από τον παραγωγό και θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτήν την διάσταση. Ο πρόεδρος. Ο κύριος Σμιθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν κοιμόμουν, να σας διαβεβαιώ. Απλώς προσπαθούσα να παρακολουθήσω τους ε, δεδάλους αυτής της εκθέσεως. Συγχαίρω τον συνάδελφο που την εκπώνησε. και την προηγούμενη Δευτέρα, όπως και πολλές άλλες φορές, έχουμε εκφράσει όλη μας την, ε, ανησυχία μας ε, για την ε, λειτουργία της αλυσίδας αφοδιασμού τροφίμων ε, είναι στιγμή νομίζω να προχωρήσουμε σε απτά ε, αποτελέσματα γιατί πολλά έχουμε πει, πολλά έχουμε δει με τις εκθέσεις αλλά ουσιαστική ε, τροποποίηση, ουσιαστικούς κανόνες στην υπόθεση αυτή δεν έχουμε δει. Ενώ έχουμε θεσπίσει με την τροπολογία μας στον προϋπολογισμό για την υπηρεσία Ασφάλεια τροφίων έχουμε εξασφαλίσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο ποσό το οποίο θα έπρεπε να πηγαίνει ακριβώς σε αυτόν τον σκοπό και ρωτώ την Επιτροπή που πήγαν τα λεφτά αυτά. Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε δεν ακούσαμε τίποτε άλλο για αποτελέσματα. Έχετε κάτι να μας πείτε από πρόοδο ως προς την ε, παρατήρηση, την δουλειά του παρατηρητηρίου για τις τιμές ε, των τροφίμων στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, δεν κοιμόμουν ούτε εγώ, αλλά δεν θέλω να πω το εξή. Για χρόνια, για πολύ καιρό συζητούμε τα θέματα αυτά, κατηγορούμε τις μεγάλες αλυσίδες, τους μεγάλους προμηθευτές, τα σούπερ μάρκετ κλπ. Ε, αλλά όπως είπε και προλύσεις, το ερώτημα είναι τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα τα έχει ο γεωργός, τα έχει ο μεταποιητής ενδεχομένως, ο παραγωγός. Ε, είναι οι τιμές, πάνω απ' όλα η σημαντική αύξηση των τιμών ε, της, ε, των καυσίμων, που συνθλίβουν τον παραγωγό και τον μεταποιητή και που βέβαια τα ανακλώνται και στη τιμή στον καταναλωτή. Έτσι λοιπόν Και όπως άλλωστε είδαμε και με την πρόσφατη κρίση στον τομέα των γαλακτοκομικών, η βραδύτητα με την οποία αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση αυτή ήταν άνευ προηγουμένου και αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την υπολογίζουν, να την λαμβάνουν υπόψη, θα πρέπει και να ανταποκρίνεται ίδια και να δρά με ταχύτητα και ε, όπως πρέπει στα προβλήματα και τις κρίσεις. Βεβαίω και θα υποστηρίξουμε ότι μέτρα είναι απαραίτητα ώστε να στηρίξουμε τα προϊόντα μας. Θα πρέπει όμως να βρούμε και την ε, χρυσή τομή μεταξύ της ασφάλειας, του δικτύου ασφαλείας όπως το ονομάζουμε, δηλαδή το κατώτατο όριο στο οποίο θα ε, πιέσουμε την αγορά. Γιατί δεν λέω ότι θα πρέπει να ελέγχουμε 100% την αγορά, αλλά θα πρέπει να την αφήσουμε και να καταρρεύσει τελείως και βεβαίως ε, ξέρουμε ότι όλοι αρέσκονται στο να διατυπώνουν ε, τις κατηγορίες τους εις βάρος των μεγάλων σούπερ μάρκετ και τα λοιπά ε, και είναι συνήθως στόχος αλλά από την άλλη και την ευελιξία έχουν και την οικονομική ισχύ έχουν και μπορούν την ώρα που μεταξύ τους αποδίδονται σε πολύ σκληρό ανταγωνισμό για να εξασφαλίσει ο καθένα το μεγαλύτερο κομμάτι τη αγορά, ταυτόχρονα μπορούν και να ρίχνουν την τιμή του γάλακτο τόσο που να είναι πιο φθηνό από το, από νερό το ίδιο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον. Άρα, πώ μπορεί ο παραγωγό να ε, διατηρήσει μια τιμή αξιοπρεπή ε, όταν το γάλα του είναι πιο ε, φτηνό από το νερό. Ο παραγωγό τελικά βγαίνει ο χαμένο από την υπόθεση αυτή, διότι ο, το σούπερ μάρκετ πιέζει το μεταποιητή, ο μεταποιητής πιέζει τον παραγωγό και τελικά κάποιος θα είναι ο χαμένος, αναγκαστικά δε, θα είναι ο παραγωγός. Για το σούπερ μάρκετ σίγουρα δεν πρόκειται να χάσει και ο μεταποιητής θα καταφέρει να βγει ίσα βάρκα, ίσα νερά, να μην χάσει δηλαδή πολλά χρήματα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Και επίσης ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος στην Ευρώπη, περιμένει από εμά. Δεν ξέρω αν την, απόφαση, την απάντηση, τη λίστα τη δώσει ένα ομπούτσμαν Ευρωπαίο ή εθνικό, δεν ξέρω τι. Αλλά πάντω ξέρουμε ότι χρειάζεται μία πλάστιγκα πάνω στην οποία να σταθμίζεται σωστά το κέρδος και το συμφέρον του παραγωγού και εκείνου ο οποίος πουλάει το προϊόν του παραγωγού αλλά και αντίστοιχα την τιμή την οποία θα ζητήσουμε από τον καταναλωτή, ώστε να είναι σωστή και η τιμή για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε την κυρία Όρβαη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ε, συμφωνήσω με τα συγχαρητήρια που εκφράστηκαν για το εξαιρετικό εγγραφό εργασία του συναδέλφου Μποβέ, επισημένοντας ότι οι πρώην σοβιετικές, κομμουνιστικές, σοσιαλιστικές αν θέλετε χώρες αντιμετωπίζουν μια ιδιάζουσα κατάσταση, όχι όλες, αλλά πάντως η δικιά μου πατρίδα η Ουγγαρία δείχνει ο μια εικόνα ακόμη πιο ε, δυσίωνη, δηλαδή η παραγωγή και η μεταπίτες σε έναν βαθμό είναι ακόμη περισσότερο στο έλεος των μεγάλων ε, αλυσίδων και των μεγάλων σούπερ μάρκετ από ό,τι στις λοιπές αγορές για τη διάθεση των προϊόντων τους. Ειδικά δε όταν έρχονται αυτές οι μεγάλες αλυσίδες για πρώτη φορά να εγκατασταθούν στη χώρα μας και όταν δεν είναι σαφής η ρόλη και η διάκριση τις ε, της ρύθμισης αγοράς, δηλαδή αρχές φοβούμενες ε, το παλαιό σοσιαλιστικό ή κομμουνιστικό παρελθόν διστάζουν να παρέμβουν στην αγορά και έτσι το αποτέλεσμα είναι και η στρέβλωση του ανταγωνισμού ισόφελος των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να κατακλείσουν την αγορά με τα προϊόντα τους στις τιμές που αυτές επιλέγουν και εις βάρος των μεταποιητών και των παραγωγών πάνω απ' όλα. Έτσι έχουμε χάσει σε μεγάλο βαθμό και τη μεταποιητική μας ε, βιομηχανία τροφίμων ε, που έχει περάσει στα χέρια των ε, ε, ξένων ε, επιχειρήσεων, ε, ιδιαίτερα η σακχαροβιομηχανία η οποία πέρασε κατευθείαν στα χέρια των ξένων, οι οποίοι αφού αγόρασαν τα εργοστάσια μετά τα έκλεισαν, γιατί αυτό που σου ενδιαφέρε μόνο ήταν να εξασφαλίσουν 100% έλεγχο της αγοράς, όχι να συνεχίσουν την παραγωγή στην Ουγγαρία. Επίσης θα ήθελα εγώ να σημειώσω ότι θα ήμουν διατεθειμένη εάν υπάρχει πρόθεση για μια μελέτη με περιπτώσεις χαρακτηριστικές για την Ουγγαρία, να σας δώσω τα απαραίτητα στοιχεία, να συμμετάσχω δηλαδή στην εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης, ώστε να έχουμε στοιχεία, στατιστικές και δεδομένα ε, από την εμπειρία της κάθε χώρας, που θα μπορούσαν πιστεύω να βοηθήσουν ε, τον ε, εισηγητή. Πιστεύω ότι μέχρι 4 Μαΐου θα μπορούσαν να έχω τέτοια στοιχεία. Are cuvântul în continuare domnul ο κύριο Ντόρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον συγγητή που εκπώνησε την έκθεση. Πιστεύω ότι είναι το όντως, το όντι, το ζήτημα αυτό ε, κεντρική σημασία για το μέλλον των γεωργών μα Σε πολλές περιφέρειες ή κράτη της Ευρώπης οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό ε, αρχές δεν μπόρεσαν να επιτελέσουν το έργο τους έναντι των μεγάλων αλυσίδων των σούπερ μάρκετ και της ανάπτυξης ολιγοπολίων από αυτές τις μεγάλες αλυσίδες με συντριπτική βέβαια ανισότητα δυνάμεως μεταξύ αυτών και των παραγωγών. Δύσκολα θα βρεθεί λύση βέβαια και η προσέγγιση που προτείνει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μου φαίνεται επαρκής ε, οι εκστρατείες καλής θέλησης ή ευαισθητοποίηση ε, για την διαχείριση των κρίσεων είναι μάλλον ευχολόγια για μένα και τίποτε περισσότερο. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση είναι η τάση στο εμπόριο να προσδιορίζονται ορισμένες φορές κανόνες που δεν έχουν βάση ε, νομοθετική. Επί παραδείγματι, στα ζητήματα της φυτοπροστασίας, ε, το εμπόριο έχει ε, επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, οι οποίοι είναι άσχετοι με αυτούς οι οποίους έχουν, έχουμε ήδη εισαγάγει εμείς στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα πρέπει πιστεύω τις εξελίξεις αυτές να τις αντιμετωπίσουμε και να τις συστήσουμε στις προσοχής Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Σταμπάιντε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να αποφύγουν τις υπεραπλουστεύσεις. Καταρχήν συγχαίρω τον εισηγητή. Για την απλοποίηση, συμφωνώ με τον κύριο Νίκολσον. Μερικές φορές ε, υπεραπλουστεύουμε τους κινδύνους των σούπερ μάρκετ. Μερικές φορές όμως ο ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ μεταξύ τους έχει και θετικούς, θετικό αντίκτυπο όπως τα ανάφερε ο κύριος Νίκολσον. Υπάρχουν πολύ δύσκολα ερωτήματα. Πώς μπορούμε να ρυθμίσουν φερπίν τις αγορές με τον κατάλληλο τρόπο ως προς την ενιαία αγορά. Παράδειγμα, η οριζόντια ενοποίηση των παραγωγών. Τι περιθώρια έχουμε. Η διαφορά είναι πολύ μικρή μεταξύ του καρτέλ από τη μια μεριά και μιας οριζόντιας ομαδοποίησης παραγωγών. Το ερώτημα αυτό δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση. Συμφωνώ με την Κομισιόν ότι ε, πολύ σημαντική είναι επίσης και η κατακόρυφη ενοποίηση. Σας ευχαριστώ κύριε Μποβέ. Όντως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης, γιατί σε εμά το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη κατακόρυφης ενοποίησης. Και λαϊκίστικα και εθνιστικά και σοβινιστικά μπορούμε να πούμε ότι οι ξένοι αγόρασαν τα εργοστάσια την βιομηχανία παραγωγής τροφίμων για να αγοράσουν την αγορά κατά κάποιο τρόπο. Σε έναν βαθμό είναι αλήθεια αυτό, αλλά οι γεωργοί εξακολουθούν να έχουν το ίδιο πρόβλημα αν ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας τροφίμων που δεν είναι συνειδιοκτήτης στο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί στην Δανία έχουμε τέσσερα σφαγεία χείρων. Και η παραγωγή είναι ιδιοκτήτες αυτών των τεσσάρων σφαγείων σε εμά, στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πέραν, άσχετο αν είναι ούγκρικο ή ξένο το σφαγείο, οι Γεωργοί δεν είναι συνειδιοκτήτες και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για μας στην Ανατολική Ευρώπη. Οι οργανώσεις παραγωγών. Μπορούμε να επικρίνουμε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά μερικέ φορές και στους αγρότες τους ίδιους και έχουμε την εμπειρία αυτή στη χώρα μας, στις νέες χώρες μέλη, οι γεωργοί δεν θέλουν να συνεταιριστούν. Εγώ είμαι γεωργικής προέλευσης και έχω, μπορώ και έχω το δικαίωμα να επικρίνω τους γεωργούς. Γιατί, τους αγρότες εννοώ. Γιατί, διότι δεν χρησιμοποιήσαμε τη δυνατότητα που παρέχουν οι οργανώσεις παραγωγών. Ο κύριος Τσόλος, ο νέος επίτροπος από τη χώρα μου, επίτροπος Γεωργίας, συγγνώμη, τόνισε την ανάγκη τοπικών αγορών. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Καλό παράδειγμα. Και πρέπει τα καλά παραδείγματα στη Γαλλία, στη Βαλονία να τα γνωρίζουμε. Ο Μάρκ Ταραμπέλα οργάνωσε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στη Βαλονία και συναντήσαμε επιτόπου τόπου φορείς οι οποίοι περνάνε την γνώση στη γεωργία όσον αφορά τις πωλήσει που θα γίνονται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Αλλά χωρίς να έχουμε ψευδεστήσεις να το αναπτύξουμε το θέμα αυτό, αλλά είναι τόσο επίδικο και τόσο ακανθώδες που πολύ δύσκολα θα βρούμε απαντήσεις. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον Έδωσα το σωστό τόνο και πιστεύω ότι επιδιώκει καλές λύσεις που μέχρι τώρα δεν έχουμε. Δυστυχώς, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στη Γερμανία είχαμε ένα σύνθημα «Ξεσηκωθείτε, έχει ξεσπάσει πόλεμος και δεν κανείς δεν πάει να πολεμήσει». Αυτό που έχω εγώ να πω ως παραλληλισμό θα ήταν ότι έχουμε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και κανείς δεν πάει να ψωνίσει. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό, γιατί έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει. Και έτσι αποφασίζει και πηγαίνει και ψωνίζει. Στα μεγάλα discount, στα φτηνά σούπερ μάρκετ, Και για να σας δώσω ένα προσωπικό παράδειγμα, η πεθερά μου έχει ένα μπακαλικάκι στο χωριό της, το οποίο τώρα, ύστερα από 70 χρόνια, κλείνει, διότι ε, ο κόσμος πάει με το αυτοκίνητο πιο μακριά στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αυτό συμβαίνει. Πάει ο κόσμος στα μεγάλα μάρκετ και ψωνίζει και όχι στο μπακάλικο του χωριού. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώ, τα προβλήματα είναι, πιστεύω, πολύ σοβαρά. Εγώ από την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στο παρελθόν ήμουνα μέλος ενός συνεταιρισμού, πάνω από, συνεταιρισμού γαλακτοκομικού με πάνω από χίλια μέλη, ίσως και οι συνάδελφοι να έχουν υπόψη τους. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα, ε, προσπαθούσαμε όσο μπορούσαμε τέλο πάντων να πουλήσουμε με, τα καλύτερα, με τις καλύτερες δυνατές ε, τιμές τα προϊόντα των ε, κτηνοτρόφων μας όσο το δυνατόν πιο καλά και ήμασταν υποχρεωμένοι λόγω του ανταγωνισμού να διατηρούμε τις τιμές μας όσο το δυνατόν ε, χαμηλά για να μπορούμε να πουλάμε. Εδώ λοιπόν με την, με την πρημοδότηση μπορούμε να έχουμε μόνο 50 εκατομμύρια μπορούμε να διαθέσουμε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της αγοράς εφόσον ο καταναλωτής δεν είναι διατεθειμένος να δώσει περισσότερα γιατί υπάρχουν ανάλογα με το τομέα της αγοράς διαφορετικές τιμές. Ε, παραδείγματι έχουμε την, φτηνή αγορά, έχουμε τα βιολογικά προϊόντα που είναι δετεθειμένος ο πελάτης να πληρώσει, ο να πληρώσει κάτι περισσότερο. Και θα πρέπει να προσέξουμε οι τιμές, οι στόχοι των τιμών που θα προσδιορίσουμε να είναι τέτοιοι ώστε να μπορούν οι παραγωγοί μας να επιβιώσουν. Διότι ο παραγωγός δεν είναι σε θέση να πιέσει το σούπερ μάρκετ. Αν μια μέρα σταματήσει να προμηθεύει ο παραγωγός το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ δεν πρόκειται καταναλωτής να καταλάβει τίποτα γιατί είναι πολύ μικρή αντιστοιχεία στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ και ο καταναλωτής δεν θα το αντιληφθεί. Επίσης στην υπόθεση του γάλακτος στα γαλακτοκομιτακά έχουμε και πολλά προβλήματα σε σχέση με μαφιώσεις και οργανώσεις και πιέσεις εις βάρος των ε, παραγωγών και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις λογικές και αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντές. Επτά είναι οι συναρφοί που έχουν στήσει το λόγο ακόμα. Πρέπει να μιλήσω. Και πρέπει να τους ζητήσω να είναι στο δυνατόν πιο σύντομοι, να μην ξεπερνούμε το 1,5 λεπτό καθένας παρακαλώ για να ακούσουμε και την Επιτροπή. Κύριος Δανέλης έχει το λόγο. Πρόεδρε, συζητάμε για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα με οικονομική και κοινωνική διάσταση που απασχολούν τον αγρότη και αντανακλούν βεβαίως τον καταναλωτή. Θα εντοπίσω την παρέμβασή μου σε ένα σημείο. Η Επιτροπή εντοπίζει σε τρεις κυρίως διαρθρωτικές αδυναμίες τις αιτίες των αποκλήσεων μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή. Στον αριθμό των μεσαζόντων που λειτουργούν στην αγροδιατροφική αλυσίδα στον τρόπο λειτουργίας του ανταγωνισμού σε κάθε στάδιο της αλυσίδας και στις ανισότητες που υπάρχουν στην διαπραγματευτική ισχύ των συμβαλωμένων μερών. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί διαφορετική προσέγγιση για κάθε διαρθρωτική αδυναμία ως εξή. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των μεσαζόντων, αυτός αναδεικνύει και το αυξημένο βάρος που πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε στην ανάπτυξη τοπικών αγορών και τοπικών δικτύων εμπορίας που μπορούν να φέρουν πιο κοντά τον παραγωγό με τον καταναλωτή και να διευκολύνουν την προσαρμογή του παραγωγού όποτε αυτή θα χρειάζεται, ενώ παράλληλα θα περιορίζουν το κόστος εμπορίας αλλά και θα προσφέρουν στον καταναλωτή καλύτερη πληροφόρηση για το προϊόν που επιλέγει. Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστική δομή στα διάφορα στάδια της αλυσίδας, πιστεύουμε ότι απαιτείται άμεσος επαναπροσδιορισμός και επανακαθορισμός εκ μέρους Επιτροπής του ρυθμιστικού πλαισίου για τις κάθετες συμφωνίες ώστε να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα το μείζον πρόβλημα τη αδιαφάνεια και τη παρεμπόδιση των απαιτούμενων προσαρμογών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, γεγονό που θα είχε άμεσα και ουσιαστικά ωφέλη τόσο για τον παραγωγό όσο βεβαίω και για τον καταναλωτή. Τέλο, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών, πιστεύουμε βεβαίω ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί ο ρόλο των παραγωγών κατά τρόπο αποτελεσματικό, γεγονό που προποθέτει την αξιολόγηση παλαιότερων σχετικών μέτρων που είχαν εφαρμοστεί και τον εντοπισμό βεβαίως και κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν αποτρέψει την απόδοση των μέτρων αυτών σύμφωνα με τις ψηλές προσδοκίες που παλιότερα είχαμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, φαίνεται ότι η γεωργική αγορά δεν είναι σε θέση να επιτελέσει το ρόλο που έχει αναλάβει. Επίσης, ο χρηματοπιστωτικός τομέας με τις τράπεζες εκεί που επιβάλλονται νέες λύσεις ή νέες αρχές επιτήρησης, αυτό που ήθελε να πράξει σύνοδος του G20. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν μετά όσα είδαμε στη γεωργική πολιτική με τους ε, διευθυντικούς μηχανισμούς. Steering δηλαδή. Ε, η παραγωγή της ε, γεωργίας αντιστοιχεί σε 15% και σε 50% και θα πρέπει ασφαλώς να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατακαιρματισμένη η αγορά και στην παραγωγή και στη μεταπίεση. Έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις ενώ ε, έχουμε ταυτόχρονα και ολιγοπόλια λίγων πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Λέγονται διάφορα λοιπόν ε, για τις ε, μεγάλες ή για τις μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά οι μικρές εκμεταλλεύσεις πώς θα υποστηριχθούν, τι θα κάνουμε για να διατηρήσουμε, να φυλάξουμε αυτό το στοιχείο που είναι το μέλλον της ε, ΚΑΠ. Ευχαριστώ κύριο Σάλβας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εδώ ένα πρόβλημα ιδιαίτερη σημασία. Γιατί και η παραγωγή και οι καταναλωτέ εξαρτώνται από αυτό. Το εισόδημα των παραγωγών εξαρτάται κατά πολύ από το πόσο θα του πληρώσει η αγορά. Και έρχονται στην αγορά μόνο μέσω αυτών των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ. Τα τελευταία χρόνια τι βλέπουμε. Μεγάλη μετατροπή, μεταβολή στην οργάνωση για πολλές αλυσίδες είτε εκ μέρους της βιομηχανίας είτε εκ μέρους των μεγάλων σούπερ μάρκετ γίνεται μεγάλη συγκέντρωση, έχουν αποκτήσει μεγάλη εξουσία. Και αυτό με στα πλαίσια κατά κάποιο τρόπο της δημόσιας παρέμβασης. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα διότι η αγορά ας πούμε οι, οι, οι σχέσεις θα πρέπει να διαμορφώνονται στην αγορά. Η αγορά είναι κάτι το θετικό, είναι κάτι το αποτελεσματικό, φέρνει διαφάνεια, πιο χαμηλές τιμές για τον αγοραστή και αμοιβή για τον παραγωγό. Αλλά αν η αγορά επέτρεπε λιγότερο ανταγωνιστικές μεθόδους ή αντιανταγωνιστικές μεθόδους και στις ε, συμβατικές σχέσεις και τις μετασυμβατικές σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να στραφούμε στις τιμές που πληρώνονται στον παραγωγό. Πρέπει να έχουμε διαφάνεια αλλά επίσης πρέπει να έχουμε και μονάδες οι οποίες να συνοδεύουν αυτή την πολύπλοκη λογική, προβληματική μάλλον, διότι οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχουν εμπειρογνώμονες. Εμείς δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό στην ελεύθερη βούληση. Πρέπει να δημιουργήσουμε εργαλεία. Πρέπει να συνοδεύουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όλα αυτά στα χέρια του ισχυρότερου. Είναι δύσκολο να φτάσουμε στον καταναλωτή αν μιλάμε συνεχώς μέσω του μεταποιητή και μέσω των αλυσίδων διανομής. Ταραμπέλα. Καταρχήν συγχαίρω και εγώ τον εισηγητή για, την, για το κείμενό του. Γιατί, γιατί πολύ σωστά πρόσθεσε δίκαιο εισόδημα για τον παραγωγό και την διατροφική και την αλυσίδα εφοδιασμού, διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Η έκθεσή του μένει βέβαια στις προτάσεις της Κομισιόν, άριστα τα, μέτρα και οι δομές, αλλά επισημαίνει και τι δεν υπάρχει. Πάμε χάρη στην παράγραφο 1 για τη διαφάνεια, πρέπει ε, να ξεχνάμε το παρατηρητήριο τιμών και περιθωρίων, ΜΑΡΖ. Μιλάμε πολύ για τη διανομή, Μιλάμε για τους παραγωγούς. Η διανομή γενικά δεν έχει προβλήματα, με εξαίρεση μερικές αλυσίδες που δεν έχουν σωστή στρατηγική, σαφή μάλλον στρατηγική, αλλά οι παραγωγοί έχουν πολλά προβλήματα. Εγώ έρχομαι από την ε, Ουγγαρία, όπου ο συνάδελφος εδώ με προσκάλεσε και διαπίστωσα ότι η αλυσίδα κόρα επεξεργάζεται ένα σύστημα όπου τα μήλα θα παράγονται επί τόπου και θα πουλούνται επί τόπου. Βραχή κύκλωμα. Παραγωγός καταναλωτής και μην ξεχνάμε τους βασικούς πρωταγωνιστές που ασκούν πίεση στο περιθώριο. Το μικρό περιθώριο του παραγωγού είναι οι μεταποιητές. Το επισημαίνει ο εισηγητής στο κεφάλαιο 2. Μιλά για την άνηση δύναμη διαπραγμάτευσης του παραγωγού και ω προ τον μεγαλέμπορο και ω προ τον μεταποιητή. Στην κρίση του γάλακτο δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Μιλήσαμε για τη διανομή, για τον παραγωγό που δεν βγαίνει. Δεν μιλάμε ποτέ για τον μεταποιητή, που είναι αυτοί που κερδίζουν περισσότερο. Και στο, στην ομάδα υψηλού επίπεδου, όταν θα έρθει το συζητήσουμε, μην ξεχάσει τον μεταποιητή, ο οποίο έχει τεράστια περιθώρια και του πιο μεγάλα από τη διανομή σήμερα. Μην του ξεχνάμε αυτού. Ουσιαστικά σε αυτό ήθελα να επιμείνω. Πρόεδρος. Ο επόμενος συνάδελφος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τον εισηγητή. Είναι ένα άκρο σημαντικό θέμα αυτό με το οποίο έχει ε, ασχοληθεί. Πρέπει να αναγνωριστεί ο παραγωγός ως παράγον της αλυσίδας και ως σημαντικός παράγον της αλυσίδας εφοδιασμού των τροφίμων. Η αλυσίδα χαρακτηρίζεται από το εξής φαινόμενο. Όπως είδαμε με το γάλα, άλλωστε πέφτουν οι τιμές και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες μέσα στην αγορά, δηλαδή αρκετή παραγωγή, τότε η τιμή φτάνει σε ένα σημείο το οποίο ε, είναι πολύ χαμηλό και αναγκάζει τον παραγωγό να παράγει ακόμη περισσότερο για να κερδίζει αρκετά. Ωραία. Καλό είναι η ελεύθερη αγορά, καλό είναι να υπάρχει ο ανταγωνισμός, αλλά πρέπει να έχει και εναλλακτικέ ο παραγωγός και πρέπει να υπάρχει και ο μηχανισμό εκείνος ο οποίος θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του παραγωγού μέσα σε αυτό το παιχνίδι θα έλεγα της ε, παραγωγής, της γεωργικής παραγωγής. Να μην είναι μόνο αντικείμενο αλλά υποκείμενο της ε, αλυσίδας παραγωγής και ε, εμπορίας. Ευχαριστώ και πρώτα τελευταία παρέμβαση ο κύριος Σάγκη. Ευχαριστώ παιδί, πολύ πρόεδρε, θα δυνατόν πιο σύντομο. Κάποιο έκανε λόγο για κατακόρυφη ολοκλήρωση και θέλω να σα αναφέρω εγώ ένα προσωπικό μου παράδειγμα, ένα ζήτημα στο οποίο έχω εγώ αναμειχθεί, με τα αυγά ελευθέρα βοσκή από το Ηνωμένο Βασίλειο, στα οποία, στην οποία υπόθεση ο συσκευαστής, η επιχείρηση συσκευασίας των αυγών έχει αναλάβει την διαπραγμάτευση εκ μέρους παραγωγού με το σούπερ μάρκετ. Τους έχει αφαιθεί δηλαδή ελεύθερο το πεδίο, έχουν πολύ μεγάλη ε, δύναμη. Ε, ελέγχουν ε, την τιμή, άλλωστε και η γυναίκα που συμμετέχει με τέτοια διαδικασία, κάθε πέμπτη γίνεται ο προσορισμός της τιμής Εάν είναι περισσότερα τα αυγά από όσα θα μπορούσε να απορροφήσει η αγορά, δεν τα ρίχνουν στην ελεύθερη αγορά, τα σπάνε, ξεχωρίζουν το ασπράδι από τον ε, κρόκο και τα καταψύχουν και μάλιστα μπορούν για μήνες, για να μην πω χρόνια να τα διατηρούν στην κατάψυξη για να τα, μεταφέρουν, για να τα επαναφέρουν μάλλον μετά στην ε, μεταπίεση όταν υπάρχει ανάγκη. Έτσι δεν επιτρέπουν να καταρρεύσει η αγορά του αυγού. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ με τα σούπερ μάρκετ είναι να έχουμε μια σήμαν σωστή, δηλαδή να μην χρειάζεται ε, να έχει αμφιβολίες ο καταναλωτής, δηλαδή να ξέρει ότι αν θέλει να πάρει αυγό από την συγκεκριμένη ε, ε, ράτσας κότα να μπορεί να το βλέπει ξεκάθαρα. Αυτό είναι μια αρρύθμιση λοιπόν ε, την οποία έχουν ε, όπως σας είπα ε, επιβάλει οι ίδιοι παράγοντες αγοράς χωρίς επιβολή άνωθεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από οποιονδήποτε άλλον ή ίδια η παραγωγή, η ίδια η παραγωγή, οι συσκευαστές, οι επιχειρήσεις συσκευασίας και οι ε, και τα σούπερ μάρκετ έχουν συμφωνήσει και έτσι διαθέτονται στην αγορά. Δεν δηλαδή, στην αγορά αυγά υψηλή ποιότητας αυγά ελευθερά βοσκή που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η ίδια η κυβέρνηση ακόμη και αν το ήθελε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενοχλητικό και απογοητευτικό το να πιέζονται προς τα κάτω οι τιμές στον παραγωγό όταν το προϊόν ταυτόχρονα στο σούπερ μάρκετ ξεκολουθεί να απόλυτε στην ίδια τιμή ή μάλιστα και σε πιο υψηλή τιμή. Η κατάσταση λοιπόν του παραγωγού στην αλυσίδα της παραγωγής βλέπουμε ότι διαρκώς επιδεινώνεται. Συνήθως τα στήλο δείχνονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες ως οι κύριοι Πέτη. Ναι, όλοι συμφωνούμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα να αναζητήσουμε συγκεκριμένες λύσεις, όλοι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λέμε ότι είναι αφέμητες οι ε, μέθοδοι που χρησιμοποιούν αυτές οι αλυσίδες και εξαντλούμε εκεί τη συζήτηση. Νομίζω ότι χρειάζεται ολοκλήρωση και ε, οριζόντια, δηλαδή μεταξύ παραγωγών αλλά και κατακόρυφη. Και επίσης υπάρχει ανάγκη για ολοκλήρωση και στην μεταποίηση, γιατί πρέπει να αντέξουμε στην πίεση των μεγάλων αλυσίδων. Εάν βραδιπορήσουμε ή εάν δεν αναλάβουμε καθόλου αυτή την πρόκληση, τότε κινδυνεύουν να δοθούν άλλες λύσεις. Θα μπορούσαμε, επί παραδείγματι, σε περίπτωση ε, αποτυχίας άλλης μεθόδου, να εισαγάγουμε κυρώσεις για τις μεγάλες αλυσίδες. Ναι, όλοι λένε νομοθετήματα, μέσα ελέγχου της αγοράς κτλ. Τι είδους μέσα όμως θέλουμε. Κυρώσεις. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις, πιστεύω. Ένα μέγιστο περιθώριο κέρδους. Κάτι μέτρα τα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολο να επιβληθούν σε χώρες όπως η δική μου τέτοιου είδους συζητήσεις δεν μπορούν καν να ξεκινήσουν ε, και μόλις πάει κανείς να πει κάτι τέτοιο αμέσως μας βάζουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της διαφάνειας. Το παρατηρητήριο μπορεί να είναι ένα στοιχείο αυτής της διαφάνειας. Αλλά δεν μπορούμε να δουλέψουμε σε μια αγορά με διαφάνεια, με σαφήνεια, αλλά δεν είναι οργανωμένη αυτή η αγορά. Άρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να δούμε πώ οργανώνουν τα διάφορα κυκλώματα με νέο μάτι. Αυτό δεν σημαίνει καρτέλ. μερικέ φορέ μπορεί να σημαίνει διαφάνεια στην ανεδιανομή των περιθωρίων κλπ. Μερικέ χώρε έχουν παρατηρήσει και η εμπειρία μα δείχνει ότι η παραγωγικότητα και το όφελος ξεκινάει από εκεί που το περιμένει κανείς η καπιταλιστική συγκέντρωση που είδαμε στα βιομηχανικά τα τελευταία χρόνια δημιούργησε νέες καταστάσεις διότι η μεγάλη συγκέντρωση ελαχιστοποιεί το κόστος αλλά προσθέτει και νέα βάρη. Δέστε πόσα νέα επαγγέλματα δημιουργήθηκαν γύρω από την αλυσίδα αυτή. Και αυτό είναι ένα βάρος, είναι ένα βάρος το, το οποίο συμπιέζει το κόστος, συμπιέζει το, το κέρδος του παραγωγού. Τι θέλω να πω. Σήμερα στην Ευρώπη έχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αντιμετωπίσουν καπιταλιστικά προβλήματα σε θέματα κληρονομιά Και υπάρχει κίνδυνος να πάνε προς τις μεγάλες αυτές δομές οι οποίε είναι σε θέση να αμύψουν τους γεωργούς με πολύ καλύτερες συνθήκες από ότι οι μεγάλες οικονομικές μονάδες. Ο κύριος Λοντέρο παρακαλώ να είναι σύντομος αν θέλει να μιλήσει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Γι' αυτό θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία. Ο κύριος στόχο του είναι να τονώσει τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Άκουσα πάρα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια από τους ε, κυρίους και κυρίες ευρωβουλευτές μετά από δύο χρόνια δουλειάς στην Κομισιόν και τρεις ανακοινώσεις για το θέμα το θέμα είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από μια πρώτη ανάγνωση του εγγράφου εργασίας βλέπουμε πολλές ενδιαφέρουσες υποδείξεις είναι φιλόδοξο κείμενο πάει πέραν από το πεδίο της ανακοίνωσης. Πάντως θα δώσουμε feedback στον εισηγητή στις ε, επόμενες μέρες. Και θα ήθελα να απαντήσω σε μια ερώτηση που ετέθη πριν από τον κύριο Σμιθ για την χρηματοδότηση κονδύλια για την Κομισιόν για ένα πιλωτικό πρόγραμμα παρατηρητήριου τιμών και περιθωρίων. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για, για την πρωτοβουλία αυτή. Είπαμε ήδη ότι όταν θα κάνουμε την ανάλυση μάλλον όταν κάνουμε την ανάλυση του παρελθόν, θεωρήσουμε ότι δεν ήταν τη στιγμή να ξεκινήσουμε με αυτή την κίνηση. Φυσικά είμαστε υπέρ ε, της πρότασης αυτής. Είμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους της Eurostat. Αυτή είναι η καταλληλότερη γι' αυτό. Δεν θέλουμε να ε, χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά του φορολογούμενου για να πάρουμε στοιχεία που ήδη υπάρχουν. Η Eurostat έχει το εργαλείο παρατήρησης των τιμών ήδη από εδώ και κάμπους μήνες δίνει στοιχεία για τις τιμές σε επίπεδο αγρόκτημα ε, μεταποιητές ε, μέχρι το εμπόριο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ την Κομισιόν. Σας θυμίζω ότι αύριο το πρωί η συνεδρία θα γίνει σε αυτή εδώ την αίθουσα. Το απόγευμα όμως θα είμαστε στην αίθουσα 2Q2 στο άλλο κτίριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE